Good morning, We will start now. Καλημέρα σας και ξεκινάμε πάλι την κοινοβουλευτική μας επιτροπή στις εργασίες της. Ξεκινάμε αμέσως με το σημείο 7. Καλημέρα σας κύριε. Με το σημείο 7 ξεκινάμε λοιπόν για εξέταση τροπολογιών για την έκθεση του κοινού συστήματος ΦΠΑ όσον αφορά την αντιμετώπιση των ε, ε, vouchers. Η κυρία Ιδικό Γκάρπερς είναι υπεύθυνη από πλευρά του ΕΛΚΑ. Έχουμε τροπολογίες τρεις που έχουν κατατεθεί και δίνω άμεσα τον λόγο τώρα στην εισηγήτρια κυρία Γκάλπες Παρακαλώ έχετε τον λόγο. Um, Σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας ήθελα να πω ευχαριστώ για τις τροπολογίες που κατατέθηκαν και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές για την επικοδομητική συνεργασία. Φορέστε, πάτε τα ακουστικά σας ε, όταν θα τα έχετε τότε και θα έχετε καθίσει για να μπορείτε να παρακολουθήσετε θα συνεχίσω. Σε συντονισμό με τους συναδέλφους μου λοιπόν έλεγα έχουμε ε, προχωρήσει σε σχέση με την πρόταση αυτή. Δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες σε σχέση με το θέμα αυτό, την έκθεση. Θα ήθελα μόνο κάποια από τα θέματα να αναφέρω σε σχέση με τις τροπολογίες. Ως αφετηρία θα ήθελα να ε, έχουμε μια συγκεκριμένη πολιτική για τα vouchers που θα είναι ενιαία και εναρμονισμένη πολιτική ώστε να αποφύγουμε οποιασδήποτε καταχρήσεις, ε, να κλείσουμε τα παραθυράκια που ενδεχόμενα υπάρχουν και να έχουμε μια πολιτική που θα επιτρέπει να αρθούμε στο ύψος ε, των περιστάσεων για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Φυσικά η φορολογική πολιτική είναι κυρίως εθνικής αρμοδιότητας θέμα από πλευράς των κρατών μελών και ε, έχουμε και την αρχή της επικουρικότητας. Έχουμε όμως και το θέμα των vouchers που χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο, ένα ευρωπαϊκό εναρμονισμένο ενιαίο πλαίσιο που θα διασφαλίζει ότι η φορολόγηση αυτών θα, είναι, ε, θα γίνεται μέσα σε ένα διαφανές πλαίσιο και θα ρυθμίζεται εξειδικευμένα. Καλωσορίζουμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η ποιότητα αυτών των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επισημαίνεται και από τις τροπολογίες που κατατέθηκαν. Ξεκινώντας με το πρώτο άρθρο, συμφωνώ πρέπει να πω με τους συναδέλφους ότι οι διαφορές όσον αφορά τα συστήματα φορολόγησης μπορεί να οδηγήσουν σε διπλή φορολόγηση πράγμα το οποίο επιβαρύνει και αποτελεί άχθος ε, για τους ε, εμπλεκόμενους στην ενιαία εσωτερική αγορά οικονομικούς συντελεστές και επιβαρύνει επίσης και το, τις διασυνοριακές ε, συναλλαγές και ανοίγει κάθε δυνατότητα πόρτες και παράθυρα για την φοροδιαφυγή. Γι' αυτό έπρεπε να έχουμε σαφείς ορισμούς. Τι ακριβώς εννοούμε με το vouchers. Και πρέπει σαφώς να καθοριστεί τη η χρήση τους για ένα σκοπό, για μία χρήση ε, εξειδικευμένα ή για πολλαπλές ε, περισσότερες ε, δυνατότητες στην χρήση τους. Όλες αυτές οι προτάσεις συμπεριλαμβάνονται στον συμβιβασμό, πρώτο συμβιβασμό, πρώτη συμβαστική τροπολογία που ελπίζω ότι θα εγκριθεί. Θέλω να τονίσω ότι η οδηγία για το ΦΠΑ πρέπει να καθιστά σαφές ότι αυτά τα vouchers θα φορολογούνται κατά την στιγμή της έκδοσης ή κατά την στιγμή της ε, εξαργύρωσής τους. Η διαφοροποίηση βασίζεται στο γεγονός ότι ε, τα στοιχεία για το ποσοστό ΦΠΑ θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ή κατά τη στιγμή της έκδοσης ή αν δεν είναι τότε ε, διαθέσιμα τότε κατά τη στιγμή της ε, εξαργύρωσής τους θα πρέπει να συμβαίνει αυτό. Και θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όλες οι συναφείς, όλα τα συναφή μέσα πληρωμών που δεν θεωρούνται ως vouchers ακριβώς κατά τη στιγμή της πώλησή τους και αυτά τα άλλα μέσα θα πρέπει επίσης να εντάσσονται υπό τους, ε, τις διατάξεις του κανονισμού αυτού σε σχέση δηλαδή με τα όσα συμβαίνουν για τα βάουτσες. Οι τροπολογίες κατέστησαν σαφές ότι συμφωνούμε ότι οι διατάξεις ΦΠΑ πρέπει να είναι σαφείς και συνεπείς όταν θα ε, μπορέσουν να φορολογηθούν με αυτόν τον τρόπο τα vouchers. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τις προτάσεις που υποβλήθηκαν από συνάδελφο για να κλείσουν τα παράθυρα όσον αφορά τη φοροδιαφυγή με αυτά τα κουπόνια. Και συμφωνώ απόλυτα με την πρόταση της συναδέλφου μας επειδή ακριβώς πρέπει να κλείσουμε τις ε, δυνατότητες ε, ε, διαφυγήσα, ή φόρο και θα πρέπει να υπάρχει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο. Γι' αυτό πρέπει να διευρύνουμε το πλαίσιο των συναλλαγών με αυτά τα κουπόνια και με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίσουμε διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Υποστηρίζω κάθε προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση. Και τώρα για, για το feedback. Αν δείτε σε σχέση με την συμβαστική πρόταση που έχει κατατεθεί, θα διαπιστώσετε ότι δέχομαι τις ε, προτάσεις ε, του κυρίου Στρατηγάκη από πλευράς των κρατών μελών θα πρέπει ταυτόχρονα αυτοί οι κανονισμοί να μπορέσουν να εφαρμοστούν και να ε, συμμορφώνονται οι πολίτες με αυτούς. Και έτσι θα μπορούμε να προσαρμόσουμε τις διατάξεις ε, των εθνικών νομοθεσιών από την 1η Ιανουαρίου 2014 και θα συμμορφωνόμεθα πλήρως ε, τότε με όλες αυτές ε, τις κανονιστικές διατάξεις από την 1η Πρώτου 2015. Πρόεδρε, νομίζω κάλυψα όλα τα ουσιαδέστερα σημεία. Προσβλέπω στις παρατηρήσεις και σχόλια των σκιωδών εισηγητών και όλων των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Thank you very much indeed. Ευχαριστώ. Κύριε κύριοι. Θα δώσω το λόγο στην σοσιαλίστρια Σκιώδη Συγήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Γκάλ για την πολύ επικοδομητική εργασία της για αυτό το τεχνικό θέμα. Μιλάμε για τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Και θα το συζητήσουμε διαμακρών σε καμιά δύο ώρες αυτό το θέμα επίσης. Και είμαι εισηγήτρια μάλιστα για αυτά τα, θέμα, για αυτά τα θέματα και θα σα παρουσιάσω τη σχετική έκθεση. Οι περισσότερε τροπολογίε λοιπόν που, που πρότεινα συνδέονται με αυτό το θέμα. Επανεξετάζοντας τι τροπολογίε, ε, προκύπτει ξεκάθαρα ότι συμφωνούμε με τι προτάσει τη Κομισιόν όλοι μα και θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό βήμα προ τα Εμπρό για να υπάρχει πλήρη ε, ουδέτερη και διαφανής ε, φορολόγηση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτω ώστε να λειτουργεί σωστά η ενιαία αγορά στην τροπολογία μου, οι τροπολογίες μου, ε, λέω ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το πεδίο εφαρμογή την ουδετερότητα και την διαφάνεια τη φορολογική μεταχείρισης των συνταλλαγών με κουπόνια. Είναι πολύ σημαντικό για την εξάλληψη ευκαιριών για φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και παράλληλα αυξάνεται η ίσπραξη του ΦΠΑ ακριβώς όπως είπε και η συγγήτρια στην παρουσίασή της, ούτως ώστε να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη σημερινή κρίση, γιατί τα εθνικά συστήματα φορολογίας είναι υποπίεση ε, και θα πρέπει να βρίσκονται πίσω και να υποστηρίζουν την πολιτική της δημοσιονομικής εξυγίανσης. Νομίζω ότι είναι καλό το έγγραφο και αυτό μαζί με τις τροπολογίες ω πακέτο πηγαίνει ακριβώς προς σωστή κατεύθυνση. Η διευκρίνηση των ορισμών είναι πολύ σημαντική γιατί πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η πρόταση τελικά θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα όλων των μορφών κουπονιών. Τέλος, ε, όταν τεθεί σε ισχύ η πρόταση, πιστεύω ότι θα έχει θετική επίπτωση στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ την εισηγήτρια ακόμα μια φορά για την ε, καλά σχεδιασμένη και προετοιμασμένη ε, έκθεση και θέλω να συζητήσουμε περαιτέρω τις τροπολογίες, τις οποίες έχουμε ήδη συζητήσει τις τελευταίες μέρες με email. Ο κύριος Γκοζές, που είναι ο εισηγητής του ΕΛΚΑ, θα πάρει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο και από όλους τους παρόντες ε, ευρωβουλευτές διαλέξετε αυτόν που μπορούσε να μιλήσει. Κυρία Γκάλπελτς, ε, σας ευχαριστούμε για τη δουλειά σας, την εκτιμούμε, σας υποστηρίζουμε σε αυτή την προσπάθειά σας για μεγαλύτερη διαφάνεια και χαίρομαι ότι οι διάφορες απόψεις συγκλίνουν για να δημιουργήσουμε μια χρήσιμη, ρεαλιστική και αποτελεσματική νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν μπορεί να πάρει το λόγο τώρα, αν θέλει να πει κάτι. Πολύ σύντομα. Ευχαριστώ την εισηγήτρια. Για την πολύ καλή συνεισφορά της, πολύ επικοδομητική, σε αυτό το πολύ τεχνικό νομοθέτημα για, την, για θέματα φορολόγησης και δείχνει ότι κατανοεί τους στόχους της Κομισιόν. Οι τροπολογίες είναι επίσης υπηρετικοδομητικές ιδίω αν λάβουμε υπόψη μας τις ημερομηνίες εφαρμογής και ακριβώς ε, συνάδει ε, με το πρόγραμμα της Ιρλανδικής Προεδρίας που σκοπό έχει να ολοκληρώσει την νομοθετική διαδικασία μέσα στο 2013 και επομένως το να έχουμε ε, ενιαίους χρόνους εφαρμογής είναι πολύ σημαντικό υπάρχει ενδυμικό πρόβλημα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 50 δισεκατομμύρια ευρώ ε, γύρω ε, κύκλο εργασιών για τις τηλεπικοινωνίες κτλ. Και η φοροδιαφυγή και οι Η νομοθεσία θα άρει τις αβεβαιότητες για τους κλάδους που προάγουν την καινοτομία. χαιρετήσουμε την πρόταση του Κοινοβουλίου και θα αντιμετωπίσουμε και τις τροπολογίες σας με πολύ θετική στάση και επικοδομητικό βλέμμα. Ευχαριστώ. Ξανά η συγγήτρια. Θέλετε ξανά το λόγο, ναι ή όχι. Όχι, δεν έχω να πω τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα. Θέλω να ευχαριστήσω τους και συζητητές, την κυρία Κλέβα, για τα καλά της λόγια, τον κύριο Γκοζές, για την ευγένειά του και να κάνω μια τελική παρατήρηση. Αν συμφωνούν και οι εισηγητές, λέω την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια συνάντηση για να οριστικοποιήσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή 3η 26 Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια θα ψηφίσουμε τον Απρίλιο. Στην Ολομέλεια λοιπόν του Απριλίου θα ψηφίσουμε αυτό το θέμα. Μπορούμε να πάμε στο επόμενο σημείο και μάλιστα θα έλεγα να πάμε στα τρία επόμενα σημεία, 8, 9, 10, οι τροπολογίες δηλαδή, για την απαλλαγή του 2011 της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της ε, ΕΣΜΑ και της ΕΙΟΠΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής δηλαδή Κινητών Αξιών και Αγορών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Στάξεων. Ο κύριος Λάγκεον ε, είναι ο εισηγητή. Έχουμε 15 τροπολογίες και για τα τρία θέματα. Πολλέ πολλές από αυτές μιλούν την, για την αύξηση α, πόρων για, για τις αρχές αυτές. Το 40% προέρχεται από τον ευρωπαϊκό Προπολογισμό και το 60% από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Ε, έτσι χρηματοδοτούνται αυτές οι υπηρεσίες. Ο κύριος Λάγκεν θα πάρει το λόγο για να μας παρουσιάσει αυτές τις τρεις εκθέσεις μαζί. Βέρνα. Ε. Ευχαριστώ πολύ. Οι τρεις αυτές ε, εκθέσεις πρόκειται για το ΕΜΠΑ, το ΕΣΜΑ και το ΙΟΠΑ. Ανήκουν στις πιο απλές, θα έλεγα, εντολές που έχω επομιστεί μέχρι σήμερα. Είναι μόνο γνωμοδοτήσεις για την Επιτροπή Προϋπολογισμού και την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού. Εδώ τα σχέδια πρέπει να τηρούνται σε συγκεκριμένα πλαίσια και γι' αυτό μόνο συγκεκριμένα θέματα έχουν ενταχθεί. Με βάση τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και τις γνωμοδοτήσεις των τριών αυτών υπηρεσιών, τα σχέδια εκθέσεων έχουν κατατεθεί και επιπλέον στις 10 Ιανουαρίου είχαμε και μια συνάντηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών με τους διευθυντές των τριών αυτών εποπτικών υπηρεσιών όπου κυρίως τρεις ε, σημαντικοί τρία σημαντικά θέματα συζητήθηκαν ως άξονες. Πρώτον, η χρηματοδότηση θεματολογικά. Χρηματοδότηση μέσα από τα κράτη-μέλη και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με μια κλίδα 60% και 40% συνολικά. Αυτό θέτει ένα πρόβλημα, διότι έχουμε αφενός και την ανεξαρτησία των τριών υπηρεσιών που πρέπει να λογοδοτούν σε σχέση με τις δράσεις τους. Και αυτό σημαίνει επίσης και ένα υψηλό βαθμό ακαμψίας, δυσκαμψίας. Γι' αυτό όλες οι διαπιστώσεις του ελεγκτικού συνεδρίου για αυτό το θεματικό θέμα πρέπει να εξεταστούν υπό την επιφύλαξη ότι η χρηματοδότηση σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα είναι άκρος προβληματική. Και γι' αυτό είχαμε και το αίτημα συναδέφων και από άλλες κοινοβουλευτικές ομάδες που διατυπώθηκε και είπαν ότι θα πρέπει να έχουμε ένα ξεχωριστό κονδύλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για όλα αυτά. Η συγχρηματοδότηση δηλαδή των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταργηθεί, πρέπει να αρθεί, ώστε να διαφυλαχθεί η ανεξαρτησία των οργάνων αυτών. Ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να διαδραματίζουν, διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο σε σχέση με τη διάθεση κονδυλίων. Όμως αυτή η κλίδα, αυτός ο επιμερισμός δημιουργεί σημαντικά προβλήματα. Το δεύτερο σημείο που επανειλημμένα αναφύεται με τις τρεις αυτές εκθέσεις, με τα τρία αυτά θέματα και γι' αυτό το συνοψίζω εδώ, είναι τι γίνεται με τα στελέχη, με τον αριθμό στελεχών όταν ξεπερνάμε κάποια όρια, τι γίνεται για την ελαστικότητα. Είπε το ελεγκτικό συνέδριο ότι υπήρχαν μια σειρά προβλημάτων για την στελέχωση, για την πρόσληψη συνεργατών, αλλά και λόγω της ε, ε, έλλειψης ε, ελαστικότητας, η ευληγησίας. Τώρα, ίσως ήταν ηθελημένο αυτό από πλευράς των κρατών των κυβερνήσεων των κρατών μελών. Αυτές οι τρεις υπηρεσίες να μην πάρουν υπερβολικές εξουσίες αυτό είναι λανθασμένη όμως προσέγγιση και τελείως ε, λάθος ε, από πολιτικής πλευράς. Γι' αυτό έχουμε και τροπολογίες που έχουν κατατεθεί σχετικά. Το τρίτο θέμα είναι τι θα γίνει με τα πλεονάσματα. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και εδώ υπάρχουν φυσικά κάποιες προτάσεις που συμπεριλαμβάνονται σε τροπολογίες που έχουν κατατεθεί. Τώρα, επισέρχομαι σύντομα σε κάποιες από αυτές ε, για την ΙΜΠΑ. Τι γίνεται εδώ. Λέγεται η κλίδα χρηματοδότησης θα πρέπει να ενταχθεί στην νομοθεσία πλαίσιο. Εκεί να ενταχθεί. Έχουμε κάποιες τροπολογίες και από πλευράς μου και από πλευράς άλλων συναδέλφων όσον αφορά ένα ξεχωριστό κονδύλιο για αυτά τα χρήματα. Μετά έχουμε και κάποιους αποσπόμενους εργαζόμενους στελέχη από τις εθνικές αρχές σε σχέση με αυτό το όργανο. Όταν όμως οι όροι και προϋποθέσεις είναι σαφείς, τότε δεν κινδυνεύει, δεν υπονομεύεται η ανεξαρτησία. Όμως για το ζήτημα της ανεξαρτησίας που τονίζεται από τα όργανα, όταν έχουμε στελέχη από εθνικές υπηρεσίες που αποσπώνται σε αυτά, δημιουργούνται πολύ συχνά τριβές όσον αφορά κάποιες ψηφοφορίες, την ψήφιση κάποιων θεμάτων. Και έχουμε και την έλλειψη ελαστικότητας, όπως προανέφερα πιο πριν, σε σχέση με τα στελέχη, όπως προσλαμβάνονται σήμερα. Έχετε τις τροπολογίες για αυτό το θέμα υπό το σημείο 8 δεν είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που προτείνονται σε σχέση με τα σημεία 9 και 10. Είναι συνολικά 15 λοιπόν τροπολογίες ε, για το θέμα ΕΜΠΑ καταρχήν. Και τώρα αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με αυτές τις ε, τροπολογίες ε, από πλευράς διατύπωσης με την κυρία Μπαμπέσκου που σε σχέση με τη ρουμανική μετάφραση υπάρχουν κάποιες ε, ε, ε, ενστάσεις. Αυτές τις τροπολογίες και αυτές τις γνωμοδοτήσεις τις αξιολογώ θετικά. Για την τροπολογία 7 του Hans Peter Martin όμως έχω ερώτηση εδώ. Προσθέτει συσσωρευτικά γραφεία εδώ με 980 τετραγωνικά μέτρα ένα εκατομμύριο 16.000 ευρώ είναι η δαπάνη και αυτό αν τα βλέπω σωστά είναι περίπου 1.000 ευρώ και βλέπουμε ε, ευρώ και παραπάνω από, για κάθε τετραγωνικό μέτρο και όταν γίνει ο σωστός υπολογισμός καταλήγουμε στα 80-90 ευρώ ανά τετραγωνικό. Ε, δεν μπορώ να κρίνω το τι γίνεται. Γνωρίζω ότι στο Λονδίνο, στο Παρίσι, στη Φραγκφούρτη είχαμε θέμα ενοικίων για τα γραφεία. Ε, τώρα συνολικά αν αυτή την τροπολογία θα την εντάξουμε, θα την δεχθούμε ή όχι, αυτό το θέμα πρέπει να το συζητήσουμε οπωσδήποτε. Μετά ο κύριος Μάρτιν έχει και την τροπολογία 9 που κατέθεσε ότι η υπηρεσία λέει δεν έχει εντολή να επιβαρύνει τα κράτη-μέλη με επιπρόσθετη γραφειοκρατική δαπάνη. Σίγουρα σωστό αυτό ως πρόταση το ερώτημα που τίθεται είναι ανήκει αυτό στην ε, έκθεση για τη χορήγηση απαλλαγή ω παρατήρηση ή όχι. Έχουμε και την τροπολογία 13 του Σβεν Γκίγκολτ που ζητεί από την υπηρεσία στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υποβάλει εξειδικευμένα πληροφορίες πριν από τον Απρίλιο 2013 να δοθούν αυτά τα τα στοιχεία γιατί δεν έχει επιτελεστεί το έργο από πλευράς της υπηρεσίας προς ικανοποίηση και ε, ευαρέσκεια του ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Αυτή η τροπολογία όμως είναι απόλυτα περιττή. Αυτό καταδεικνύει ότι η συνάδελφος Γκίγκολ δεν ασχολήθηκε με αυτό το θέμα σε βάθος γιατί πρώτον με την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου έχουν δοθεί γνωμοδοτήσεις σχετικά. Είχαμε και τη δημόσια ακρόαση όπου εξειδικευμένα απαντήθηκε αυτό το ερώτημα, αυτό το ζήτημα. Και τρίτον και εγώ και άλλοι είχαμε επιπρόσθετες διαβουλεύσεις και συζητήσεις που κατέληξαν σε προτάσεις σε σχέση με τη δική μου ίδια ε, έκθεση, το σχέδιο έκθεσής μου. Είναι λοιπόν περιττή λογοδιάρεια αυτή από πλευρά του συναδέλφου, απορρίπτω ο αυτές τις προτάσεις του. Με όλα τα άλλα μπορώ να τα δεχθώ τα υπόλοιπα όπου εδώ ε- ετέθη το θέμα σε σχέση με τον κύριο Μάρτιν, δεν βρίσκεται όμως εδώ. Αν αυτά τα ακριβή αριθμητικά στοιχεία τα οποία αναφέρει σε σχέση με την συσσόρευση, την αθρηστική τους αυτή παρουσίαση αν αληθεύουν και μπορούν έτσι να γίνουν δεκτά ή όχι. Απομένει αυτό το ερώτημα σε σχέση με την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Και για τη 13 του κυρίου Γκίγκολ που, απορρίπτει, που απορρίπτω όλες τις άλλες τις δέχομαι. Αυτά είχα να πω σε σχέση με το σημείο της, για το ΕΜΠΑ. Πρόεδρος, σα ευχαριστούμε πολύ κύριε Λάγκεν. Τώρα θα δώσουμε τον λόγο στη συνέχεια στην κυρία Φερέιρα, εξ ονόματο της σοσιαλιστική Ομάδας, παρακαλώ. Πολύ σας ευχαριστώ κύριε Λάγκεν. Εμείς πιστεύουμε ότι γενικά στοχεύουμε στις ίδιε κατευθύνσει, όπως η τοποθέτηση που παρουσιάστηκε από εσά μόλι πριν. Θεωρούμε και εμεί με άλλα λόγια ότι οι υπηρεσίες αντιμετωπίζουν νέα καθήκοντα και καθήκοντα απόλυτης υψηλών απαιτήσεων και δεν είναι δυνατόν να λείπουν τα υπαρκή οικονομικά στοιχεία και να μην μπορούν να κάνουν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους όπως προβλέπεται. Πρέπει κάτι να κάνουμε λοιπόν και για τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ε, τα κονδύλια με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο απαιτεί ένα επαρκές επίπεδο, ένα ικανοποιητικό επίπεδο αμοιβών. Και Επίσης για τα στελέχη, τους υπαλλήλους, πρέπει να είναι σε θέση οι υπάλληλοι να καλύψουν πολύμορφα τον πολυσχηδή χαρακτήρα και από τεχνικής πλευράς των καθηκόντων που επομίζονται. Ως προς όλα αυτά λοιπόν η κύρια ανησυχία μας, το κύριο μέλημά μας είναι να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα αυτών των εποπτικών αρχών. Τούτων λεχθέντων τώρα, εμείς πιστεύουμε ότι θα ήταν σημαντικό να είχαμε αξιολόγηση με σοβαρό τρόπο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της χρηματοδότησης ε, για να δούμε τι μπορεί να γίνει σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τις ανάγκες τους. Θα ήταν η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να διασφαλιστεί η απόλυτη ανεξαρτησία αυτών των θεσμικών οργάνων και να αντιμετωπιστεί η οποιαδήποτε αβεβαιότητα ώστε να έχουν την δυνατότητα να ε, ε, κάνουν τα καθήκοντά τους όπως πρέπει. Και στη μεταβατική αυτή φάση που η εποπτεία πρέπει να διασφαλιστεί και να εδρεωθεί καλά, μέσα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, πώς να το πω, θα έδινα θα ήθελα να διασφαλίσουμε περισσότερο την ανεξαρτησία, την προβλεψιμότητα και βεβαιότητα για τις δράσεις αυτών των οργάνων. Αυτές είναι οι κυρίες παρατηρήσεις μας. Ευχαριστούμε για το πνεύμα συνεργασίας του κυρίου Λάγκεν και των συναδέρφων που εμπλέκονται σε σχέση με αυτήν την έκθεση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Εσμή, εκ μέρου ε, τη Άλντε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δυστυχώ έχασα το πρώτο τμήμα της παρέμβασης του κύριου Λάγκε, αλλά δεν θα συμφωνήσω με τον Σβάνγκη, τουλάχιστον ελπίζω ότι δεν θα είμαι στο ίδιο μικρό Ευχαριστώ τον κύριο Λάγκεν και τα όσα ακούστηκαν δείχνουν ότι είμαστε πάνω κάτω στην ίδια πλευρά. Στην ομάδα μας, όπως ξέρετε, ζητάμε και επιμένουμε αυτοί, αυτές οι αρχές και η εποπτεία τους ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ενισχυθεί. Αυτό βεβαίω είναι περίπλοκο. εάν δεν υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για τις αρχές αυτές και αυτό αντικατοπτρίζεται νομίζω και σε όλες τις τροπολογίες. Ο κύριος Λάγγεν ανέφερε αυτές τις τροπολογίες σε όλες τις εκθέσεις. δάλος βεβαίως θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και η ομάδα μας προσπάθησε να συγχωνεύσει όλες αυτές τις αρχές σε μία. Νομίζουμε ότι αυτό θα είναι πιο αποτελεσματικό και για το μέλλον αυτό ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση. Ένα επιπλέον επιχείρημα είναι ότι αν δώσουμε επιπλέον καθήκοντα σε αυτές τις αρχές, όπως και έχουμε πράξει, σε οδηγίες και κανονισμούς, για τους ε, οίκους αξιολόγηση και ούτω καθεξής, αν το κάνουμε αυτό, βεβαίως είναι σκόπιμο να τους παρέχουμε και την κατάλληλη χρηματοδότηση. Η συνάδελφος που κάθεται δίπλα μου θα είναι υπεύθυνη για τον προπολογισμό. Όλοι ξέρουμε αυτή τη συζήτηση και είναι επίκαιρο το θέμα. Ακόμα και αν εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί στις δαπάνες μας. Αλλά αν αναθέτουμε περαιτέρω καθήκοντα, πρέπει να έχουμε και επιπλέον χρηματοδότηση. Όπως είπε και ο κύριος Λάγκεν, έχουμε κάποιες κοινέ ε, τροπολογίες και σε όλες τις εκθέσεις. Πολύ ωφέλιμο και χρήσιμο αυτό. Και τώρα μήπως θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές ε, στις ε, χρηματοδοτικές διευθετήσεις. Αυτό βεβαίως δεν μπορούσαμε να το εξετάσουμε. Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί. Τι συμβαίνει με τις αμοιβέ, ε, τα υπέρ και τα κατά της αξιοποίησής τους. και πώς συνδέεται αυτό με την ανεξαρτησία τους, ε, που για μένα είναι εξαιρετικά σημαντική. Αν δηλαδή λαμβάνουμε έσοδα από αυτούς τους οποίους ελέγχουμε, πώς ε, ε, αυτό επηρεάζει την ανεξαρτησία της αρχής. Είναι σημαντικό θέμα και ίσως χρειαζόμαστε νέες, πιο σύγχρονες μεθόδους Πρέπει λοιπόν να τα εξετάσουμε και είδα ότι και η Λίσα Φερέιρα έχει καταθέσει τροπολογίε ε, προ αυτή την κατεύθυνση. Οφέλιμο αυτό. Θα μείνω εδώ. Δεν θα είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση, πιστεύω. Και στο τέλος θα υπάρχει ευρεία πλειοψηφία. Ευχαριστώ, κύριε Σμιτ. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των πρασίνων της GUE του ECR. Α, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Περιμένουμε ακόμα τον καφέ ή λίγο νερό, αλλά γενικά συμφωνούμε με, την, με τις εκθέσεις του κυρίου Λάγκεν. Να είμαστε δίκαιοι. Εγώ δεν είμαι και ειδικό γιατί υπεύθυνη είναι η κυρία Σουισβόρν και δεν βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Βάσει όμως ε, ορισμένων παρατηρήσεων μπορώ να σας πω να σας υπενθυμίσω την έκθεση Ashley Fox για τον προπολογισμό του 2012. Εμείς ε, ψηφίσαμε ότι ε, εφόσον θα μπορούσαν να υπάρξουν ε, εξοικονομήσεις, αν και υπήρχαν κάποιες εξοικονομήσεις που δεν μπορούσαν να γίνουν, υπήρχαν και κάποιες ασυνέπειες στις δαπάνες από τον ESA. Και θα ήθελα εδώ να το επισημάνω για παράδειγμα στις μεμονωμένες γραμμές προπολογισμού. Από πλευράς μας λοιπόν θα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ό,τι αφορά τις δαπάνες που συνδέονται με τον ESA. Και είμαστε σχεδόν σίγουροι ότι ευθυγραμμιζόμαστε με τη θέση του κ. Λάγκεν. Αυτά τα ολίγα για μια έκθεση για την οποία εγώ δεν είμαι υπεύθυνο. Ευχαριστώ κύριε Στρέικερ. Ζητώ συγγνώμη πριν που δεν σα έδωσα το λόγο. Κύριε Λάγκε, παρακαλώ. Ε. ναι, σα ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται να φοβάται ο συνάδελφο Σμιτ ότι θα αντιμετωπιστεί ισοπεδωτικά η πρότασή του. Έχουμε αυτέ τι τροπολογίε. Ευχαριστώ του Σοσιαλδημοκράτε για την υποστήριξη όλες τις τροπολογίες με εξαίρεση την τροπολογία 13 που τη θεωρώ απόλυτα περίτη μπορούμε να τις θέσουμε σε ψήφιση. Το θέμα είναι το αν η τελευταία τροπολογία η 15 υπενθυμίζει ότι πρέπει να έχουμε 100% κοινοτική χρηματοδότηση αυτών των υπηρεσιών, μήπως αυτό μέσω άλλων τροπολογιών καλύπτεται ήδη ίσως. Όχι ε, από πλευράς της διατύπωσης, αλλά σε σχέση με την ουσία με τη 14 την 11. Αυτό είναι το μόνο ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Θα πρότεινα να περάσουμε τώρα στο, στο ε, έγγραφο αξιολόγησης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Λάγκαν. Θα πάρει τον λόγο ο κύριος Μαντ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο Βέρνερ Λάγκαν έκανε ήδη μια σύνοψη που παρουσίασε για αυτό το θέμα. Αυτό το οποίο διαπιστώνω είναι ότι ο Όλε δεν έχει μια ισοπεδωτική αξιολόγηση σε σχέση με αυτό έχουμε σε σχέση με αυτά τα θέματα και θετική ε, ας το πω έτσι, επίδοση του κύριου Όλε Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Χαίρομαι ότι υπάρχει ομοφωνία με τους ε, σοσιαλδημοκράτες. Η κυρία Φερέρα κατέθεσε τροπολογίες που στοχεύουν προς την ίδια κατεύθυνση. Το ερώτημά μου είναι σαφές Βέρνερ. Αν μπορούμε να το καταφέρουμε να έχουμε ένα κονδύλιο ξεχωριστό, αυτή είναι η βάση που χρειαζόμαστε για να δουλέψουμε σωστά. Δεύτερον, όσον αφορά την εξοικονόμηση, δεν είναι μόνο θέμα στελεχών υπαλλήλων, είναι θέμα δυνατότητα τα διαθέσιμα αυτά στελέχη να ξέρουν ότι υπάρχει ένα νέο λειτουργικό πλαίσιο το οποίο μπορεί και πρέπει να εφαρμοστεί χωρίς να πρέπει νέα στελέχη να προσληφθούν διότι παντού λένε να εξοικονομείτε, να εξοικονομείτε, να εξοικονομείτε στο τέλος πρέπει να έχουμε δυνατότητα ώστε να λειτουργήσουν σωστά τα αναγκαία ε, επίπεδα, ενδιάμεσα επίπεδα γι' αυτό να πούμε το αν κάτι είναι υπερβολικά δαπανηρό ή όχι δεν είναι τόσο απλό να κρυθεί. Σημαντικό είναι όταν έχουμε πρόσθετα καθήκοντα τα οποία θέλουμε να καλυφθούν και πρέπει να καλυφθούν πρέπει να δούμε αν μπορούμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι είσαστε σε θέση να κάνετε αυτή τη δουλειά. Νομίζω είναι σε θέση να το κάνουν αυτό. Τίθεται το ερώτημα ότι πρέπει ή μπορούμε ή δεν μπορούμε να έχουμε πρόσθετο ε, προσωπικό. Να δούμε από τις ανάγκες που υπάρχουν μπορούμε με ένα ευσύνοπτο τρόπο να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σε σχέση με την κατάσταση που ε, παρουσιάζεται σήμερα από την ΕΜΠΑ. Αυτό είναι το ερώτημα αν μπορούμε σε σχέση με τις ε, διάφορες ανάγκες να πούμε ότι χρειάζεται αυτό ή όχι. Στο τέλος δεν χρειάζεται κάποιο συμβούλιο να μας πούν περικόπτω με τα κονδύλια και να δείτε στο τέλος τι θα καταφέρετε. Πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε λειτουργικό επίπεδο που θα διασφαλίζεται και γι' αυτό θα δώσει το καλό παράδειγμα η Ευρωπαϊκή Εποπτεία Τραπεζών. Αυτό είναι το θέμα. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας ευχαριστώ κύριε Μαν. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην κυρία Γένσεν. Παρακαλώ κυρία Γένσεν. Εισηγήτρια της Επιτροπής ε, Ελέγχου Προπολογισμών. Ο Όλε Σμιτ είναι ο εισηγητή, σκιώδη εισηγητής για αυτό το θέμα. Εγώ ασχολούμαι το προπολογισμό του 2014. Και το θέμα της χρηματοδότησης αυτών των ε, αρχών υπηρεσιών είναι κάτι για το 2014 πρέπει να το δούμε. Ευχαριστώ τον κύριο Λάγκεν και όλου όσου ασχολήθηκαν για την έκθεση. Είναι καλή βάση εργασίας για τους μελλοντικού προπολογισμού. Είχαμε συναντήσεις με αυτές τις αρχές και υπάρχει ακριβώς αυτό το θέμα της χρηματοδότησης από τα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη δεν μπορούν να πληρώσουν. Δεν έχουν το πλεόνασμα, θέλουν να πληρώσουν σε φάσεις, σε δόσεις. Αυτό δημιουργεί περιττή γραφειοκρατία και υπάρχει το θέμα της ανεξαρτησίας βέβαια που είναι πολύ κρίσιμο. Πρέπει να αλλάξουμε όμως τον κανονισμό για να αλλάξει κάτι τέτοιο. Η Επιτροπή σας έχει την... Συγγνώμη, η Επιτροπή των Προπολογισμών έχει την αρμοδιότητα, όχι εγώ, αλλά προτείναμε να το εξετάσουμε στην Επιτροπή Προπολογισμών. Κάτι που ανέφερε και ο Λε Σμιτ τώρα. Είναι μήπω θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί, να χρηματοδοθούν και οι τρει αυτέ υπηρεσίε εν μέρη αποτέλει στο μέλλον. Ίσως θα κοιτάξουμε, θα πρέπει να έχουμε μία μεταβατική φάση χρηματοδότηση από τον κοινωτικό προπολογισμό και συνεχεία ενδεχόμενη χρηματοδότηση από τέλη. Αλλά μην ξεχνάτε και τι γίνεται με τα κράτη-μέλη που πληρώνουν για τη λειτουργία και τα λειτουργικά έξοδα αυτών των εποπτικών αρχών. Το βασικό είναι να έχουμε διαφανείς αρχές ε, για το πώς θα διαμορφωθούν αυτά τα τέλη. Αν δείτε έναν άλλο τομέα όπου χρησιμοποιούνται τέτοια τέλη από υπηρεσίες, υπάρχει πρόβλημα διαφάνειας. Θα πρέπει να τα κάνουμε εδώ καλύτερα τα πράγματα. Το, το τελευταίο που θέλω να πω ότι αυτές οι υπηρεσίες παραπονιούνται για τα οργανογράμματά τους. Σας συστήνω λοιπόν όταν περάσετε στην πραγματική διαδικασία προϋπολογισμού να κοιτάξετε τα οργανογράμματα αυτών των υπηρεσιών. Μερικές φορές δεν είναι το πρόβλημα τα χρήματα, δεν έχουν το σωστό οργανόγραμμα και την ευελιξία που χρειάζεται, ούτω ώστε να φέρουν ε, και να προσλάβουν τους κατάλληλους ανθρώπους για τις συγκεκριμένες θέσεις. Πάντως, σας ευχαριστώ κύριε Λάγκεν για αυτές τις εκθέσεις, είναι θαυμάσιες και συμφωνώ απόλυτα με τα όσα προτείνετε και θα προσπαθήσουμε και εμείς από πλευρά μας να συνεχίσουμε, να πάρουμε τη σκητάλη. Ευχαριστώ κύριε Γένσεν. Ο κύριος ε, Λάγκεν μπορεί να δευτερολο... θέλει να δευτερολογήσει, δεν ξέρω. Ευχαριστώ για την υποστήριξη. Το θέμα της ερώτησης ε, του κυρίου Τόμας Μάν σε σχέση με την κυρία Γιάννη αμέσως να το απαντήσω στην, στο επόμενο θέμα που θα συζητήσουμε για το ΕΣΜΑ. Για το ΕΣΜΑ έχουμε τις περισσότερες τροπολογίες που είναι ταυτόσιμες αλλά έχουν διαφορετική αρρύθμιση. Επί της ουσίας όμως είναι θα έλεγα σε μεγάλο βαθμό ταυτόσιμες. Και επιπρόσθετα στο ΕΣΜΑ δεν έχουμε επιπρόσθετες τροπολογίες που να έχουν κατατεθεί γι' αυτό. Όμως, εδώ έχουμε το θέμα της χρηματοδότησης ε, των ε, ε, δαπανών, την χρηματοδότηση από προϋπολογισμό των κρατών μελών. Αυτό τίθεται ως θέμα. Αφενός με το ερώτημα τι θα γίνει με τα πλεονάσματα. Δεύτερον, με το θέμα ή με την τοποθέτηση ότι οι εθνικές αρχές θέλουν να ανακτήσουν το δυνατόν μεγαλύτερα κονδύλια. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου με άλλα λόγια για το αν η υπηρεσία έχει μεγαλύτερες δαπάνες και πρέπει πιο εντατικά να εργάζεται. Σύμφωνα με την άποψη του ΕΣΜΑ, αυτό η ανάκτηση κονδυλίων από τα κράτη-μέλη και τους προπολογισμού τους ε, έχει επιπτώσεις σε σχέση με τις δαπάνες και την κάλυψη των δαπανών της, ε, του ΕΣΜΑ. Γι' αυτό υπάρχει το αίτημα μεγαλύτερη της ελαστικότητας για τη διάθεση και χρήση των κονδυλίων. Κατέστη σαφές κατά τη διάρκεια της εξέτασης του θέματος αυτού ότι στην ε, φάση εγκατάστασης, ε, εγκαθίδρυσης αυτής της υπηρεσίας αυτό το θέμα δεν είναι ίσονος σημασία. Γι' αυτό έχω και την τροπολογία μου 11 που κατέθεσα για το σημείο 8 που την αρχική μου γνωμοδότηση κάπως την απαμβλύνει παρακαλεί το ελεγκτικό συνέδριο τα προσκόμματα που υπάρχουν ή τα εμπόδια που υπάρχουν να τα εξετάσει ιδιαίτερα εξειδικευμένα για την πρώτη φάση αυτή την, της έναρξης, την ενακτήρια φάση λειτουργίας του ΕΣΜΑ και να δούμε τι θα γίνει για τη χρηματοδότηση. Το αποφασιστικό θέμα είναι αυτό το οποίο επαρκώς καλύπτεται από τις τροπολογίες θα έλεγα. Κατά τα άλλα, τι έχουμε. Σε μεγάλο βαθμό έχουμε ταυτόσιμες τροπολογίες, το είπα ήδη από κάποιους συναδέφους απόλυτα ταυτόσιμες τροπολογίες με τις άλλες για τα άλλα όργανα, τα άλλα θεσμικά όργανα που κατατέθηκαν προηγούμενα. Για την ΕΣΜΑ δεν έχουμε πρόσθετες τροπολογίες. Για τη ΓΙΟΠΑΜΑ είχαμε, ναι. Thank you very much indeed. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λάγκεν. Κύριε Οδησηγητά, θέλετε να απαντήσετε να σχολιάσετε τις τροπολογίες για την ΕΣΜΑ, αλλιώς ε, να δώσω το λόγο και πάλι στον κύριο Λάγκεν για τις τροπολογίες ΕΙΟΠΑ. Ε, Μάλιστα. Για αυτές τις τροπολογίες ε, ακριβώς στον ίδιο βαθμό έχουμε μια υποεγκαθίδρυση υπηρεσία, ένα θεσμικό όργανο που βρίσκεται στην φάση ανάπτυξης του. Και έτσι σε σχέση με την κυρία Φερέρα εδώ, όπως για την ΕΜΠΑ πιο πριν, ενώ όχι για την ΑΙΟΠΑ. Σωστό αυτό. Για την ΑΙΟΠΑ τι βλέπουμε ότι έχουμε. Έχουμε μια τροποποίηση που είναι γλωσσικού αποκλειστικά χαρακτήρα. Κατά τα άλλα οι τροπολογίες είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό ταυτόσιμες. Τώρα η ακρόαση τι οδήγησε να αντιληφθούμε. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ΑΙΟΠΑ ιδιαίτερα υπό το πρίσμα των εσωτερικών οικονομικών ελέγχων καταλήγει στο να πει ότι θα ελέγχονται και από τις εθνικές αρχές. Και αυτό είναι σχετικά πολύ για το 60% των ελέγχων αυτών. Και το πρόγραμμα εργασίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την χρηματοδότηση που θα διασφαλιστεί. Θα έχει και νέα καθήκοντα που θα αναλάβει η ΑΙΟΠΑ. Το ίδιο λοιπόν ισχύει όπως και για τις άλλες εθνικές αρχές. Στο τέλος τέλος δηλαδή του επόμενου οικονομικού έτους που θα ολοκληρωθεί θα πρέπει να ξαναπροβληματιστούμε και να δούμε πώς ενδεχόμενα μέσω πρωτοβουλειών τη χρηματοδότηση αυτή θα μπορέσουμε να την τροποποιήσουμε ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Αυτό είναι τελικά το ερώτημα. Με παρόμοιο τρόπο τίθεται για την ΑΙΟΠΑ όπως και για τα άλλα όργανα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λάγκεν. Οι συγητέ, σκιώδει θέλετε να σχολιάσετε, κύριε Μάν, παρακαλώ. Ε, Ουσιαστικά μόνο το θέμα και στη δική σου έκθεση Βέρνερ για το θέμα της εποπτείας των αξιογράφων, των χρεογράφων. Έχουμε και την τροπολογία Μάρτιν και τώρα εδώ για την ΑΙΟΠΑ την υπαριθμόν οκτώ τροπολογία. Πάντα το ίδιο δηλαδή. Διαπιστώνεται ότι δεν έχει εντολή ε, η υπηρεσία αυτή να επιβαρύνει τα κράτη-μέλη με πρόσθετη γραφειοκρατική επιβάρυνση. Δεν πρέπει να δημιουργείται αυτή η γραφειοκρατική επιβάρυνση. Αυτό μου θυμίζει πάντα τη φρικτή κατήχηση των ε, ε, κυριακάτικων κατηχήσεων που ακούμε και δεν γίνονται φαίνεται τα πράγματα σωστά. Δεν επαρκούν όλα αυτά. Είναι, περιτεύουν αυτές οι τροπολογίες. Θέλουμε να οδηγήσουμε στο αποτέλεσμα να λειτουργούν αποτελεσματικά και να μην δημιουργείται γραφειοκρατική επιβάρυνση. Είναι και οι δύο θα έλεγα περιτές. Ποια είναι η δική σου άποψη. Τι λες εσύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάν. Κύριε Λάγκεν παρακαλώ. Να απαντήσω. Σε αυτό το θέμα έχω κάπως διχασμένη άποψη. Έχω μακρά πείρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δείχνει ότι τα ευρωπαϊκά όργανα ε, δεν είναι πάντα ικανά να επιλύουν αυτά τα προβλήματα όπως θα έπρεπε. Ενώ θα μπορούσε να γίνεται αυτό. Το να υπάρξει λοιπόν μια ανεξάρτητη εντολή, διασφάλιση ανεξαρτησίας όπως διασφαλίζεται μέσω εντολής, να μην ανοίξουν πόρτες και παράθυρα όμως ε, να ε, υπάρχουν εξαιρέσει. Θεωρώ ότι είναι σωστό το αίτημα. Θα ξαναπροβληματιστώ να δω για την τροπολογία 8 του κυρίου Μάρτιν αν θα προτείνω ξεχωριστή ψηφοφορία ώστε ένα μέρος των επιχειρημάτων να μπορέσει να καλυφθεί τουλάχιστον με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Ας σταματήσουμε εδώ λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Σας υπενθυμίζω ότι ε, στην Επιτροπή θα ψηφίσουμε στις 25 Φεβρουαρίου στην Ίκον και στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού στις 9 Μαρτίου. Και τέλος στην Ολομέλεια η ψηφοφορία θα γίνει ή τον Απρίλιο ή τον Μάιο. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της μέρης σας διάταξης, σημείο 14 γιατί όπως ξέρετε έχει αναβληθεί η ψηφοφορία. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 14. Έκθεση λοιπόν για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων. Η συγκέντρια είναι η κυρία Κλέβα από τους σοσιαλιστές. Να της δώσω το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε περίπου 1-3 ευρώ δημοσίων χρημάτων χάνεται κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της φοροδιαφυγής και της φοροαπαλλαγής, φοροαποφυγής. Και αυτό περίπου ανέρχεται σε 2.000 ε, ευρώ κόστος για κάθε Ευρωπαίο πολίτη. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους λοιπόν, ιδίως ε, εν καιρό κρίσης όπου κάθε ευρώ που μπορούμε να συλλέξουμε πρέπει να το συλλέγουμε και να το δαπανούμε καταλήλως. Αλλά χάνουμε περίπου όσα χρήματα ε, ξοδεύει κάθε κράτος μέλος ε, στην υγεία, για παράδειγμα, αυτό αποτελεί και μια απειλή για το κοινωνικό ε, πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ό,τι αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες. Απειλή και για την ενιαία αγορά και σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα και την δικαιοσύνη στα φορολογικά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η απώλεια εσόδων συνεχώς αυξάνει το επίπεδο ελλημάτων και χρεών ε, των κρατών μελών. Εξαιτία τη ε, φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή, ε, πόροι που αλλιώ θα πήγαιναν σε επενδύσει, στην ανάπτυξη και την απασχόληση, χάνονται μέσα σε αυτέ τι φορολογικέ τρύπε, αν θέλετε. Κανένας δεν θα διαφωνήσει μαζί μου ότι αυτά τα προβλήματα είναι πραγματικά πολύ στην Ευρώπη και πρέπει πραγματικά κάτι να κάνουμε. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και είμαι σίγουρη ότι και σήμερα η συζήτηση θα είναι γόνιμη. Κατανοώ ότι τα κράτη-μέλη διατηρούν την αρμοδιότητα σε ό,τι αφορά το φορολογικό του σύστημα και η δράση σε εθνικό επίπεδο είναι πολύ σημαντική. Όμω στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία με την διασυνοριακή φύση τη ε, φοροδιαφυγή, ε, τα μονομερή εθνικά μέτρα από μόνα του δεν μπορούν να έχουν ε, τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γι' αυτό και στην έκθεσή μου ζητώ την σύσταση ενός ε, πολύ συγκεκριμένου τεκμηριωμένου και ολοκληρωμένου συστήματος και στρατηγικής ε, σε τη φορολογική πολιτική ε, που θα εστιάζει και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό και στο διεθνές επίπεδο. Θεωρώ ότι έχει έρθει η ώρα να, να τολμήσουμε. Δεν θέλω να επαναλάβω το σχέδιο δράσης που προτείνει η Επιτροπή, που καλύπτει κυρίως ε, τεχνικά θέματα. Το σχέδιο δράσης ε, κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, όμως θα ήθελα περαιτέρω νομοθετικέ προτάσεις από την Επιτροπή και ε, να εκδηλωθεί και μια ισχυρή πολιτική βούληση από τα κράτη-μέλη. Στην έκθεση ζητώ να υπάρχει ε, ο κύριος στόχος να, μειωθεί κατά 50% αυτό το φορολογικό κενό μέχρι το 2020. Ένας τέτοιος φιλόδοξος ε, στόχος θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να, έχουν περισσότερα έσοδα από φόρους χωρίς να αυξήσουν τους φορολογικούς συντελεστές. Με αυτόν τον στόχο δεν θα ε, αυξηθούν και τα δημόσια έσοδα μόνο από ε, τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, αλλά θα έχουμε και άμεσα αποτελέσματα. Θα οδηγήσει στην σταθεροποίηση των χρηματοοικονομικών αγορών μέσω της σημαντικής μείωσης της διαθέσιμης ρευστότητας ε, για τις ε, χρηματοοικονομικές συναλλαγές που δεν συνδέονται με την οικονομική δραστηριότητα. Όλα θα ξεκινήσουν από τα κράτη-μέλη εκείνα θα πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους και να επισέλθουν σε σοβαρές διαπραγματεύσει για να κλείσουν όλες τις ανοιχτές νομοθετικές προτάσεις σε ζητήματα φοροδιαφυγής και φοροποφυγής. Πρώτα απ' όλα έχουμε την αναθεώρηση της ε, ε, οδηγίας περί καταθέσεων είναι σημαντικό τα κράτη-μέλη να ολοκληρώσουν τις μονομερείς τους ε, διαπραγματεύσεις και να δώσουν το πράσινο φως στην Επιτροπή για να γίνει εκείνη το ε, σώμα φορέας που θα διαπραγματεύεται τέτοια ζητήματα με, με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην έκθεση ε, αναφέρω ένα κατάλογο δραστηριοτήτων με, την οποία, με τις οποίες μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή αλλά και τη φοροαποφυγή που είναι νόμιμη βεβαίως, όμως ε, με αυτή την στρεβλή ε, αξιοποίηση του φορολογικού συστήματος έχουμε ακόμα περισσότερες ε, δυσμενείς επιπτώσεις από ότι στην φοροδιαφυγή. Μετά, μεγάλες επιχειρήσεις τεχνητά μεταφέρουν τα κέρδη τους για να ελαχιστοποιήσουν τον φορολογικό τους συντελεστή και να μειώσουν το φορολογητέο τους εισόδημα. Ε, πρέπει να έχουμε μία τεκμηριωμένη σειρά επιχειρημάτων ε, για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πράγματα και προβλήματα. Ε, ενέργειες πρέπει να αναβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα, τραπεζική αδειοδότηση η οποία θα ανακαλείται σε τέτοιες περιπτώσεις μετά μια κοινή φορολογική, επιχειρηματική φορολογική βάση. Ε, να επικαιροποιήσουμε το πεδίο εφαρμογή ε, τη οδηγία περικαταθέσεων, ε, να αναθεωρήσουμε το πλαίσιο για τι διασυνοριακέ επιχειρήσει και να ενισχύσουμε τα μητρώα επιχειρήσεων ή e trust. Υπάρχουν και άλλες ενέργειες όπως είναι η αυστηρότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής μέσω ποινική δίωξης ε, και αντιμετώπιση του προβλήματος ε, του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ε, ηλεκτρονικού οικονομικού εγκλήματος. Άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα στην έκθεσή μου είναι η φορολογική παράδειση. Ο που είναι ηγετική δύναμη σε αυτό τον τομέα ε, έχει εδώ και χρόνια καταρτήσει το δικό του κατάλογο των φορολογικών παραδείσων και αυτός ο κατάλογος σήμερα είναι άδειος. Αυτό δείχνει από μόνο του πόσο αναποτελεσματικές ήταν οι εργασίες σε αυτόν τον τομέα. Κατά τη γνώμη μου, δεν, τίποτα δεν πρέπει να σταματά, σταματά την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει τον ηγετικό ρόλο με ένα νέο ε, ε, ξεκάθαρο ορισμό βάσει διεθνών προτύπων αλλά και ε, εγκαθιδρυμένων κριτηρίων μπορούμε και θα έπρεπε να, να καθορίσουμε λοιπόν κριτήρια και μέτρα που πρέπει να αναλυφθούν για να ε, τα διευθετήσουμε όλα αυτά. Χρειαζόμαστε μια κοινή αντιμετώπιση απέναντι στους φορολογικούς παραδείσους και βεβαίως έχουμε και το σχέδιο δράσης της Επιτροπής αλλά πρέπει να δημιουργήσουμε και μια δική μας ευρωπαϊκή ε, μαύρη λίστα. Τέλος, να σχολιάσω και τις δεσμεύσεις Γερμανών, Γάλλων και του Γερμανού, Γάλλου και Βρετανού ε, Υπουργού Οικονομικών την προηγούμενη εβδομάδα στην ομάδα στη συνάντηση του G20 στη Μόσχα. Όλοι μαζί είπαν ότι η φοροαποφυγή είναι άδικη και ότι οι πολυεθνικές θα πρέπει να σταματήσουν ε, να καταχρώνται τις παγκοσμιοποίησεις και να πληρώνουν ε, το μερίδιο που τους αναλογεί. Όλοι επίση είπαν ότι πρέπει να αλλάξουμε την νομοθεσία και η αποφυγή να καταστεί παράνομη. Βεβαίως και χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι υπάρχει πολιτική βούληση, τουλάχιστον να αυξάνεται αυτή. Και δεν πρέπει να αφήσουμε τέτοιε ευκαιρίε να πάνε χαμένε. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες ε, αναλαμβάνουν δεσμεύσει λοιπόν να καταπολεμήσουν τη φοροαποφυγή, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι υπουργοί εμποδίζουν όλες αυτές τις ε, συναφείς προτάσεις στο Συμβούλιο. Φαίνεται ότι δεν έχουν ε, τη δέσμευση να συντονίσουν τη συλλογική δράση σε επίπεδο G20 και γι' αυτό οφείλουμε να διασφαλίσουμε ε, οι ίδιες δεσμεύσεις να αναλαμβάνονται και σε ό,τι αφορά τις δικές μας ε, προτάσεις. Ουσιαστικά τους δίνουμε αυτό που μας ζητούν, προτάσεις για δράση. Και νομίζω και ελπίζω ότι σε αυτή την Επιτροπή θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση και προσβλέπω στην ε, συνεργασία μου με τους ασκιώδεις συζητητές εδώ και σε άλλες συνεδριάσεις. Ευχαριστώ κυρία Κλέβα από το ΕΛΚ. Θα σας δώσω το λόγο, μισό λεπτό. Πρώτα να δώσω το λόγο στους σκιώδεις συζητητές και μετά στον κύριο Λάγκεν. Πρέπει να σεβαστούμε τη σειρά με την οποία παίρνουν το λόγο οι διάφοροι ομιλητέ. Κυρία Πικάνεν, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη θαυμάσια προσπάθειά της. Είναι καλή βάση για να προωθήσουμε περαιτέρω αυτό το θέμα. Είναι μια καλή πρωτοβουλία της ε, Επιτροπής μας. Και καλό θα ήταν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το αντιμετωπίσει. Υπάρχει τεράστια τεράστιο πρόβλημα φοροδιαφυγής και ε, φοροαποφυγής και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα μαζί. Έχοντας υπόψη μας και το στόχο της δημοσιονομικής εξυγίασης και τις ανάγκες του ενωσιακού προϋπολογισμού και τον εθνικό προϋπολογισμών. Μισή, ε, ορισμένες εκτιμήσεις λένε ότι ο, τα ποσά που φοροδιαφεύγουν είναι, ανέρχονται στο 1 σε εκατομμύριο. Αλλά είναι πολύ σημαντικό και για τις κοινωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι οι πολίτες και οι φορολογούμενοι μας δεν μπορούν να πιστέψουν σε ένα σύστημα όπου οι πλούσιοι κάνουν ότι θέλουν στην πραγματικότητα, ενώ κάποιοι άλλοι φέρουν το βάρος μόνοι τους Νομίζω ότι και από αυτή τη σκοπιά είναι ακόμα πιο σημαντικό να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Θα σταθώ σε κάποια από τα θέματα πολύ σημαντικά, που είναι πιο σημαντικά, γιατί το θέμα είναι πολύ ευρύ. Η ο φορολογικός ανταγωνισμός είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά αυτό που είναι άδικο είναι αυτά τα συστήματα ε, επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού σε ορισμένα κράτη-μέλη και πώς γίνεται κατάχρηση του συστήματος. Ξεκινάμε με αυτόν τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, με τη, με τη διάθεση για φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Ε, υπάρχουν μια σειρά από εργαλεία και όλα μαζί πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Σε κάτι που θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο, που λέει και η έκθεση. Είναι η δουλειά που κάνει το G20 και ο Αναφέρει η έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει πιο ενεργό ρόλο με συγκεκριμένες προτάσεις σε διεθνές επίπεδο για αυτά τα θέματα. Θα υποβάλω προς αυτήν την κατεύθυνση κάποιες τροπολογίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις που έχουμε. Ποινικές συμφωνίες για τα θέματα της φοροαποφυγής. Και είναι η ποινική διάσταση του θέματος, μάλλον, για αυτό το θέμα. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα πολύ συγκεκριμένα και γι' αυτό θα υποβάλω ε, τροπολογίες. Πώς μπορούμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την υπάρχουσα νομοθεσία σε διάφορα φόρουμ, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Καλά παραδείγματα είναι ε, η έκθεση για τον εταιρικό φόρο η συνεργασία, η υποχρεωτική συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορολογικών αρχών και μου αρέσει η ιδέα ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα την νομοθεσία και τον κανονισμό για τα χρηματοοικονομικά. Παραδείγματος χάρη, να αντιμετωπίσουμε τις το θέμα των αδειών που έχουν ε, οι τράπεζες, τράπεζες οι οποίες δεν συνεργάζονται και δεν αντιμετωπίζουν τη φοροδιαφυγή. Εν πάση περιπτώσει δεν κάνουν τίποτα για την εμποδίσουν. Επίσης ε, υπάρχει και οδηγία για την καταπολέμηση του ξεπλήματος του χρήματος. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και αυτή. Το δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω είναι η διεθνή συνεργασία αλλά και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ένας ε, ευρωπαϊκός ε, αριθμο, φορολογικός αριθμός είναι πολύ σημαντικός. Ε, η οδηγία για, τα, για τους τόκους και τα δικαιώματα. Επίσης, ένας, μια ευρωπαϊκή μαύρη λίστα για τους φορολογικούς παραδείσους. Οι συμβάσεις για τη διπλή φορολόγηση πρέπει να αντιμετωπιστούν και να αρθούν αυτές οι συμβάσεις με αυτές οι χώρες που θεωρούνται φορολογική παράδειση και να ανανεωθούν με ένα τέτοιο τρόπο που όπως λέει και η Κομισιόν να εμποδίζουμε την διπλή φόρο Φυσικά η διπλή φορολόγηση είναι ε, παράνομη, αλλά χρησιμοποιούν αυτή την νομοθεσία με αδικαιολόγητο τρόπο αυτοί που θέλουν να φοροδιαφύγουν. Εν πάση περιπτώσει, έχω μια καλή ευκαιρία εδώ στο Κοινοβούλιο, ούτω ώστε να υποβάλουμε ένα εκτεταμένο κατάλογο στο Συμβούλιο και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και που θα αντιμετωπίζει και το θέμα της αρχής, τα θέματα των αρχών, αλλά και το συγκεκριμένο δράσεων που πρέπει να προωθήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύο φαινόμενα της φοροδιαφυγής και της φοροποφυγής. Ευχαριστώ κυρία Πικάνεν. Ο κύριος Κυλακάκης από τους φιλελεύθερους και συγγνώμη που σκότωσα το όνομά σας. <laughs> Όχι, ωραία το είπατε. Έχω ακούσει και χειρότερα από τα δικά σας. Συμφωνώ με τους ε, προλαλήσαντες και τον, την εισηγήτρια ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και είναι πολύ καλή έκθεση κιόλα. Το θέμα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και φορολογικής απάτης είναι σημαντικό. Όχι μόνο αν το δούμε από τη σκοπιά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γιατί δεν μπορούμε να έχουμε μια σωστή φορολογική ένωση όταν έχουμε διαφορετικά επίπεδα φορολογικής απάτης σε διάφορες χώρες. Γιατί η φοροδιαφυγή, όταν είναι ευρεία και εκτεταμένη, επηρεάζει την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγείων σε μια χώρα. Οι εξαγωγείς συνήθως δεν έχουν τη δυνατότητα να φοροδιαφύγουν. Γιατί εξάγουν εκτός της χώρας. Όταν υπάρχει μεγάλη φοροδιαφυγή, υποσκάπτεται λοιπόν η ανταγωνιστικότητα των περιφερειακών οικονομιών. Αν κοιτάξουμε και το φορολογικό χάσμα, και αν υποτεθεί ότι επιλύουμε αυτό το πρόβλημα και δεν υπάρχει αυτό το φορολογικό χάσμα πια. Όχι μόνο. Όχι μόνο αυξάνει το βιωτικό επίπεδο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δημιουργούμε και ένα σοσιαλιστικό κράτος, αν δεν μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές. Η διαφορά εδώ είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί προς τη φοροδιαφυγή και να αντιμετωπίσουμε το θέμα των φορολογικών παραδείσων και αυτό και τα κρατη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επιδιώξουν ενεργά. Δεν θα πρέπει όμως όλα αυτά τα έσοδα να επιστρέφουν στα εθνικά ταμεία. Γιατί αν όλοι αυτοί οι φόροι αυξήσουν το βαθμό της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία, τότε δεν θα είμαστε ανταγωνιστικοί ως Ένωση εν γέννη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση και για την, ε, το φορολογικό ανταγωνισμό μέσα στην Ευρωζώνη. Δεν έχουμε εργαλεία, ούτως ώστε οι διάφορες οικονομίες να αντιμετωπίσουν το θέμα της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι διάφορες οικονομίες της ε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να προσαρμόσουν την νομισματική του πολιτική, γιατί όλε οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ίδια νομισματική πολιτική, δεν μπορούν να παίξουν με τις ε, φορολογικέ του πολιτικές, γιατί τώρα κινούμαστε προς ε, μια πολύ έντονη δημοσιονομική εξυγίαση, χωρίς ελλείμματα κτλ. Επομένως, πώς θα μπορέσουν οι περιφερειακές οικονομίες, οι οικονομίες της περιφέρειας να κρατήσουν ανταγωνιστικότητά τους εάν σε κάποια φάση δεν έχουν αρκετή έρευνα, τεχνολογία και καινοτομία και δεν μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους ε, με άλλου τρόπου. Θα πρέπει να έχουν χαμηλότερου φόρου, ούτω ώστε να μπορούν να μείνουν στο ίδιο επίπεδο. Τώρα, σε διάφορε χώρε έχουμε ανεργία 27%. Πώ μπορούν να προσελκύσουν επενδύσει, Και έχουμε και διαφορετικά επιτόκια. Τρία έχουμε διαφορά τριών-τεσσάρων ποσοστιαίων μονάδων. Γιατί ο πυρήνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και η περιφέρεια έχουν τέτοιε διαφορέ. Πώ θα, θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσει αν δεν έχουμε χαμηλότερου φόρου. Θα πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε τη δυνατότητα για φορολογική, φορολογικό ανταγωνισμό παράλληλα με την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ευχαριστώ κύριε Σκυλακάκη. Ευχαριστούμε κύριε Σκυλακάκη. Ευχαριστώ Θεοδόρα. Θα λάβει τον λόγο για τους πράσινους τώρα. Ο κύριος Σέικαουτ, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και πιθανότατα δεν θα προσπαθήσω εγώ να προφέρω το όνομά σας, διότι θα ακουστεί ακόμα χειρότερα. Έχουμε προβλήματα με την προφορά αυτών των ονομάτων μας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ από πλευρά εισηγητού για αυτό το πρώτο σχέδιο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των φοροπαραδείσων είναι σαφέ ότι στο γενικό επίπεδο όλοι συμφωνούμε με την φοροδιαφυγή και τους φορολογικούς παραδείσους ότι θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα εξάπαντος. Αυτό που βλέπω να απουσιάζει στην έκθεση είναι μια σαφή τοποθέτηση ότι ένα από τα προβλήματα είναι το βέτο για κάθε κράτος μέλος, για κάθε φορολογικό θέμα. Αυτό είναι ένα από τα μείζωνα προβλήματα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη φάση. Αφενός, από τη μια πλευρά, διαρκώς συζητούμε όλο και περαιτέρω μέτρα λιτότητα και δημοσιονομική πειθαρχία, λιγότερε δαπάνε από πλευρά των κυβερνήσεων. Από την άλλη πλευρά, εξακολουθούμε να επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να ανταγωνίζονται στα φορολογικά θέματα, οδηγώντα σε μικρότερα εισοδήματα, λιγότερα έσοδα στα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να πει στι κυβερνήσει πρέπει και πάλι να, να δαπανάτε λιγότερα χρήματα. Βλέπουμε στα θέματα φορολόγηση δεν κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την FDT για την ε, ομάδα που θα έπρεπε να είναι μπρος-μπρος να δούμε τι γίνεται σε σχέση με την νομοθεσία. Όλα αυτά τροχοπεδούνται στο Συμβούλιο για θέματα φορολόγησης Και όταν έχουμε θέματα φοροδιαφυγής φοροαπάτη, φοροπαραδείσων, θα πρέπει να διασφαλιστεί θα έχει μια πιο ενδυναμωμένη, ενισχυμένη θέση η Ευρωπαϊκή Ένωση και να ακολουθήσει την κοινοτική μέθοδο και να γίνει αντιληπτό ότι μια και ο Κάμερον ούτως ή άλλως ε, έχει ξεπεράσει αυτό το όριο, εμείς στο Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε σαφέστατοι και να πούμε ότι εμείς ως Ευρωβουλή εργαζόμαστε για μια αλλαγή της συνθήκης για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν κοινοτικέ μέθοδοι που θα υιοθετούνται για τέτοιου είδους ε, θέματα φορολόγησης. Και γι' αυτό λοιπόν με τις τοπολογίες αυτές θέλουμε να ενδυναμώσουμε αυτές τις ε, κατευθύνσεις. Για άλλα θέματα θεωρούμε ότι επιπτώσεις της φοροδιαφυγής ε, στα αναπτυσσόμενα κράτη ως ε, συνιστόσα πρέπει και αυτή να συμπεριληφθεί στην έκθεση. Η φοροδιαφυγή πλήττει ιδιαίτερα τι αναπτυσσόμενε χώρε, διότι έχουν και προβλήματα όσον αφορά αυτού του είδου τον ανταγωνισμό. Θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτών των φορολογικών θεμάτων για αυτά τα κράτη, λαμβάνοντα υπόψη ιδιαίτερα τι επιπτώσει για τα αναπτυσσόμενα κράτη. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να καλύψω και στην έκθεση αυτή πρέπει να ενδυναμωθεί είναι το ότι Επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πιο αυστηρή σε σχέση με τον ορισμό του TSD φοροπαράδεισος, φορολογικός παράδεισος. Καθώς είμαι και Ολλανδός πρέπει να πω μάλιστα η Ολλανδία είναι φορολογικός παράδεισος. Και θα ήταν τρομερό αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθυστερεί για να υποβάλει κάποια πρόταση για ε, κάποιο υποφελή ορισμό για το TST φοροπαράδεισος ξέρουμε ότι δεν είναι υπέρ, ιδιαίτερα υπέρ οι Ολλανδοί υπέρ ενός τέτοιου αυστηρού ορισμού διότι αμέσως θα ταυτοποιηθούν, θα ταυτιστούν ως φοροπαράδεισος. Όμως ε, γνωρίζω ότι από πλευράς ε, του ε, Ολλανδικού Κοινοβουλίου υπάρχει διατύπωση που απαγορεύει την χρήση του, του όρου φοροπαράδεισος. Δεν ξέρω αν αυτό είναι παράνομο τώρα αυτό που προτείνω σε σχέση με το Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Όντας στις Βρυξέλλες όμως θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά ότι θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ορισμό των φοροπαραδείσων. Να είμαστε πιο απαιτητικοί και αυστηροί. Εκείνο που θα ήθελα να ληφθεί υπόψη και για ένα άλλο Ολλανδικό ζήτημα είναι να δείξουμε ότι η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή επιδεινώνει την ε, οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Ας δούμε τους λόγους που δείχνουν ότι μεταθέτουν την έδρα εγκατάσταση στους ε, εταιρείε ε, από την Πορτογαλία στην Ολλανδία. Λόγω φοροδιαφυγής, λόγω φοροανταγωνισμού πρέπει αυτά τα θέματα να ενταχθούν επίσης στην έκθεση αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχω πολλούς συμμάχους στην ίδια μου τη χώρα με αυτά τα οποία λέω, αλλά εγώ γι' αυτό έχω εκλεγεί εδώ. Να είμαστε έντιμοι και ακέραιοι και τα θέματα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής είναι θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν οπωσδήποτε. Ευχαριστώ για τη συνεργασία για αυτά. Σας ευχαριστώ κύριε Κάουτ. Τώρα ο κύριος Στάγεκ, εξ των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούγοντας την εξέλιξη αυτής της συζήτησης προσεκτικά και παρακολουθώντας αυτά τα οποία αναφέρθηκαν, πρέπει να πω ότι είχα προετοιμάσει πάρα πολλά σχόλια από πλευράς μου για αυτή την έκθεση. Έχοντας ακούσει όμως το μέρος της συζήτησης που ε, εξελίχθηκε με αυτόν τον τρόπο, Αναδιατύπωσα απόλυτα τις παρατηρήσεις μου και τα σχόλιά μου. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που άκουσα και ακούω εδώ και άκουσα σήμερα. Η πρώτη μου παρατήρηση κιόλας κιόλας αφορά αυτό ίσως σας δείξει ότι είναι κάτι ξεχωριστό. Όμως θα ήθελα να ρωτήσω πόσοι από αυτούς που βρίσκονται εδώ γύρω από αυτό το, τραπέζι έχουν αναλάβει καθήκοντα να είναι επικεφαλής επιχειρήσεων και πόσοι από εμά έχουν πείρα, είχαν ευκαιρία να καταναλώσουν κάποια προϊόντα που αφορούν ε, φορολογικούς κώδικες και ε, προϊόντα φορολογικών αρχών και υπηρεσιών. Εγώ είχα τέτοια πείρα, είχα την επιχείρησή μου και γνωρίζω από πρώτο χέρι περί τίνος πρόκειται και τι σημαίνει με όλα αυτά να έχει κανείς να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα να ε, εκτελέσει, να κάνει κάποιο έμβασμα, να στείλει χρήματα, να περιμένει κάποιο έμβασμα και να αναμένει οι αρμόδιες φορολογικές αρχές να ε, εγκρίνουν ή να διαφυβάσουν ε, κάποια τέτοια θέματα, να θα διεκπαιρεώσουν σε σχέση με τους επιχειρηματίες. Είναι λοιπόν και λυπούμε, είναι τόσο εύκολο να πει κανείς ότι απολεσθέντα ε, έσοδα ή χρήματα θα μπορούσαν με άλλο τρόπο να έχουν χρησιμοποιηθεί. Είναι εύκολο καμιά φορά να χειραγωγήσει κανείς, να εξοραίσει, να χειραγωγήσει την ίδια την πραγματικότητα και να τη φέρει στα μέτρα του. Συγγνώμη, διαφωνώ. Πάντα θα είμαι στην πλευρά ο σύμμαχος των απλών πολιτών που επομίζονται καθημερινά κινδύνους με το να έχουν μια επιχείρηση υπευθύνη τους. Αν δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι αυτοί που θα μπορούν να επομιστούν και να αντιμετωπίσουν αυτούς τους κινδύνους. Κανείς από εμά δεν θα βρισκόταν στη θέση του εδώ, γύρω από αυτό το τραπέζι σήμερα. Και λυπούμε για αυτή την διαφωνία ή ένσταση από πλευράς μου ή την, ε, την οργισμένη αυτή παρατήρησή μου θα πρέπει να ηρεμήσουν περισσότερο ίσως ε, τα πνεύματα και οι τόνοι. Μετά από τη συζήτηση αυτή, όντας μέσα στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης, το κύριο ερώτημα είναι γιατί οι επιχειρήσεις φοροαποφεύγουν ή κάποιες από αυτές ε, ανακατευθύνουν τα κεφάλαιά τους ώστε η ροή αυτών των κεφαλαίων να καταλήγει σε φοροπαραδείσους. Αυτό είναι το σωστά διατυπωμένο ερώτημα δεν είναι αναγκαίο να ε, φιλοσοφήσει κανείς επί παντός του επιστητού για επιχειρήσεις, αλλά να ρωτήσει γιατί κάνουν αυτά τα πράγματα οι επιχειρήσεις. Απάντηση, η λόγοι είναι απλή. Υψηλή φορολογία και υπερβολική φόρη, υπερβολικά περίπλοκοι φορολογικοί κώδικες και απόλυτα κατανόητες ε, φορολογικές ε, αρμοδιότητες και εξουσίες και υπερβολικοί περιορισμοί όσον αφορά τους επιχειρηματίες και τη δράση τους. Πρέπει να τα πούμε όλα αυτά και να τα κατονομάσουμε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι, οι πολίτες, και εγώ δεν είμαι στο πλευρό εκείνων που χρησιμοποιούν το μέσο της φοροαπάτης ε, και μάλιστα και καθημερινά και κανένας δεν μπορεί να ε, δεχθεί κάτι τέτοιο αλλά η φοροαποφυγή που είναι κάτι το οποίο δεν έχει αναφερθεί κιόλα καθόλου σε αυτή την έκθεση εγώ θεωρώ ότι είναι υπό την εξή μορφή Θέλουμε ή δεν θέλουμε να υπάρχουν νόμιμες δραστηριότητες σε συγκεκριμένα πλαίσια. Διότι αυτή η φοροδιαφυγή ή η φοροαποφυγή είναι άμεσο αποτέλεσμα υπερβολικά ε, περίπλοκων, ακατανόητων και δυσλειτουργικών κανόνων και κανονισμών. Και αν όλα αυτά στο ευρωπαϊκό επίπεδο μετατεθούν με τον ίδιο τρόπο η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί σημαντικά καθόλου θα εξακολουθήσουμε χωρίς καμιά αμφιβολία να έχουμε την ίδια περίπλοκη κατάσταση, την ίδια δυσνόητη κατάσταση, χωρίς να μπορεί να είναι λειτουργική. Και μια τέτοια κατάσταση θα καταλήξει σε ροές κεφαλαίων προς τους φορολογικούς παραδείσους. Ας κάνουμε και δεκάδες οποιασδήποτε ε, διατάξεις, αυτό θα συνεχιστεί αν παραμείνουν τα πράγματα έτσι λοιπόν. Λυπούμε, οι τροπολογίες μου εξακολουθούν να υφίστανται Αυτές ήταν οι αναδιατυπωμένες μου παρατηρήσεις. Οι τροπολογίες μου λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση ευθυγραμμίζονται. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much indeed, Mr. and I because... Ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη, νόμιζα ότι είχατε ολοκληρώσει. Εκ μέρου τη ΓΚΟΕ να δώσω το λόγο στον κύριο Χέντελ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τώρα με βάση αυτά που ανέφερε ο προλαλής σας πρέπει και εγώ να κάνω μια εκπροημίου παρατήρηση. Μέχρι την έναρξη της κοινοβουλευτική μου εντολής είχα μια μικρομεσαία επιχείρηση που ήμουν επικεφαλής αυτής. Κάποιος μπορεί ίσως να έχει πλαγεί ότι ένας της αριστεράς είχε μια τέτοια επιχείρηση. Όμως να σας πω, σε μία πτυχή των παρατηρήσεών σας κύριε αν συμφωνώ. Δεν χαίρεται κανείς ποτέ όταν παίρνει ραβασάκια από την εφορία. Σπάνια χαίρεται κανείς για κάτι τέτοιο. Δεν θα κατέληγα όμως την ιδέα για υποτιθέμενη υπερβολική ρύθμιση φορολογικών θεμάτων να σκεφτώ να καταλήξω να στείλω χρήματα σε ένα φοροπαράδεισο ή να φοροδιαφύγω ή να φοροαποφύγω διότι εδώ πρόκειται για κοινωνικές δαπάνες που για κοινωνική χρήση πρέπει να χρησιμοποιούνται με αυτά τα κονδύλια και όταν φοροδιαφεύγει κανείς δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και για ένα δημοκρατικό όργανο σε σχέση με, ε, ιδιαίτερα με έναν προϋπολογισμό που συντάσσεται, όμως οι φόροι είναι κοινωνική ευθύνη και όποιος φοροαποφεύγει και φοροδιαφεύγει δεν το κάνει, σπάνια το κάνει από ό,τι γνωρίζω εγώ για τους λόγους ότι είναι περίπλοκοι λέει οι κανόνες και οι κανονισμοί. Το κάνει λόγω απουσίας κοινωνικής συνείδησης και συνειδητοποίησης και λόγω εγκληματικής ε, πρόθεσης να φοροδιαφύγει. Λοιπόν, για την πρόθεση που μπορεί να είναι καλή αλλά με πολλούς δισταγμούς και επιφυλάξεις. Και βλέπουμε εδώ θα πρέπει να υπάρξει λέει αξιολόγηση και αυτό γίνεται επί σειρά ετών και πού θα καταλήξουμε και, στους δύο, και στα δύο επίπεδα και στη φοροδιαφυγή και στη φοροαπάτη κατεπηγόντως χρειάζονται βελτιώσεις και πρέπει να βελτιωθούν τα πράγματα. Πρόσφατα ο ΣΑ με μια δραματική έκθεση επισημαίνει ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και προτείνει μέτρα να ληφθούν και προαναγγέλλονται αυτά τα μέτρα για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ήδη σήμερα είναι κάποια τέτοια μέτρα εφικτό να υιοθετηθούν. Κάποιες από αυτές τις προτάσεις εμπεριέχονται και στην έκθεση της εισηγήτριας. Πολλές από τις προτάσεις αυτές μπορούμε να τις υποστηρίξουμε. Μας ικανοποίησε ιδιαίτερα το αίτημα προς τα κράτη-μέλη και συμπεριλαμβάνεται αυτό όλες οι συμφωνίες διπλής φορολόγησης ε, με όλες τις χώρες ε, να καταργηθούν όσον αφορά τη διαφάνεια για παράδειγμα που πρέπει να διαφυλαχθεί και εκείνους που δεν τη διαφυλάσσουν με αυτόν τον τρόπο. Θα υποβάλουμε και περαιτέρω προτάσεις ώστε σήμερα, εδώ και τώρα ήδη, στον τομέα της φοροαποφυγής και αφοροαπάτης να δυσχερανθούν πόρτες και παράθυρα ως διάβλη και να έχουμε την δυνατότητα για τον, την μέθοδο υπολογισμού να είμαστε αποτελεσματικότεροι. Και τα τραπεζικά ιδρύματα από μη συνεργάσιμες χώρες πρέπει να αφαιρεθεί η άδεια ε, συναλλαγών από αυτά τα ιδρύματα. Και δεν είναι δυνατόν να, ε, να συνεχίζουν να φοροδιαφεύγουν κάποιοι με αυτούς τους τρόπους. Θεωρούμε ότι τα ευρωπαϊκά ε, χρηματοπιστατικά ιδρύματα όταν έχουν ε, ιδρύματα ε, θυγατρικές ε, σε χώρες που δεν, μπορούν, δεν θέλουν να συνεργαστούν πρέπει με τον ίδιο τρόπο να προχωρήσουμε για όσες χώρες δεν συνεργάζονται με την Ευρώπη θα πρέπει από τα κράτη-μέλη να υπάρχει φορολόγηση επί της πηγής με 50% εξάπαντος. Αυτές είναι προτάσεις που συνεισφέρουν στο να βελτιωθεί η έκθεση περαιτέρω. Ελπίζουμε στην υποστήριξή σας. Όπως η συγγήτρια πολύ σωστά διαπιστώνει, είναι σκανδαλώδης η κατάσταση ότι έχουμε ένα δις ευρώ μέσω της φοροαπάτης και της φοροδιαφυγής. Κάτι πρέπει να κάνουμε επιτέλους και πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως, άμεσα, εδώ και τώρα. Αυτό θα ήθελα να πω με αυτή την παρέμβασή μου. Και αντίθετα με τη θέση του προλαλήσαντος από την Άλντε, δεν είναι δυνατόν περαιτέρω ευρωπαϊκοί φόροι να οδηγούν σε περαιτέρω ανταγωνισμό, φοροανταγωνισμό και dumping, φορολογικό dumping. Όλα αυτά αποβαίνουν εις βάρος των κρατών μελών και εις βάρος των κοινωνιών αυτών των κρατών μελών μας, των πολιτών τους. Αυτό πρέπει να σταματήσει και να σκεφτούμε επιτέλους για ένα ελάχιστο επίπεδο φορολόγησης ευρωπαϊκού χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Χέντερ. Στον κατάλογο έχουμε την κυρία Ιντφελτ, Γκάπες Μακάρθη και Γκουλάρ. Υπάρχει άλλος που θα ήθελε να παρέμβει σε αυτό τον συμπληρώνω σε αυτόν τον κατάλογο. Η κυρία Ιντφέλτ παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να απαντήσω στα όσα είπε ο κύριος Στάκεκ. Βεβαίω ε, και οι φορολόγηση θα πρέπει να είναι δίκαιοι, τα συστήματα φορολόγηση και συλλογή φόρων πρέπει να είναι αποτελεσματικά, να αποφεύγεται γραφειοκρατία. Όμω δεν νομίζω ότι θέλατε κι εσεί να πείτε ότι οι εκατομμυριούχοι και οι δισεκατομμυριούχοι που διοχετεύουν τα χρήματά του από την Ελλάδα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία, ότι αυτό είναι ένδειξη επιχειρηματικότητας. Βεβαίως και όχι. Και αν ε, δούμε και τις ε, αντιδράσεις, στη χώρα μου για παράδειγμα, κατέστη σαφέ ότι τα μέλη τη ε, βασιλική οικογένεια είχαν χρήματα σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις Βρετανικές νήσους, βεβαίως και ο κόσμος δεν και ιδιαίτερα. Εξορισμού, αν κάποιο θέλει να βάλει τα χρήματά του σε ένα τραπεζικό λογαριασμό κάπου που δεν μπορούν να φτάσουν ε, οι αρχέ, εξορισμού κάποιο δεν έχει χρήματα. Αν, αν κάποιο δεν έχει χρήματα, μάλλον δεν χρειάζεται να τα στείλει σε κάποιο φοροπαράδεισο. Αυτοί που έχουν λοιπόν εξορισμού θα φοροδιαφύγουν και θα φοροαποφύγουν. Θα ήθελα εδώ να θίξω δύο συγκεκριμένα ζητήματα. Ε, το ένα αφορά την ε, ε, ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαφάνεια, που είναι κύριο σημείο σε αυτή τη διαδικασία. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι σημαντική, αλλά θα πρέπει και να ρυθμίζεται. Πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών, ποιος έχει πρόσβαση στις πληροφορίες και για ποιου σκοπού μπορεί να, να χρησιμοποιούνται οι πληροφορίε αυτέ. Βλέπουμε ότι πολλέ φορέ αυτό δεν ρυθμίζεται. Κάποιοι είπαν ότι ε, υπάρχουν δύο χώρε που μπλοκάρουν όλε τι ε, συμφωνίε και αυτό οδηγεί στο ότι οι ευρωπαϊκέ κυβερνήσει εμποδίζουν και λειτουργούν ω τροχοπέδι σε αυτήν την ανταλλαγή πληροφοριών. Πρέπει να μπει πολύ πιο ψηλά στην ατζέντα αυτό το θέμα. Άλλο ζήτημα που θέλω να θίξω εδώ Υπάρχει κεφάλαιο για τη διεθνή συνεργασία. Ανησυχώ ιδιαίτερω για το ΦΑΤΚΑ, ε, ε τον νόμο, τον ΙΠΑ που θα τεθεί σε ισχύ φέτος το καλοκαίρι, που θέτει τεράστιο βάρος ε, στα χρηματοοικονομικά ιδρύματα που λειτουργούν στις ε, ΙΠΑ. Και είναι λοιπόν υποχρεωμένα αυτά τα ιδρύματα να παράσχουν πληροφορίε για του Αμερικανού πολίτε ή Αμερικανικέ αρχέ που έχουν τραπεζικού λογαριασμού στην Ευρώπη. Αυτό αποτελεί παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Και ε, κάποια κράτη-μέλη έχουν συνάψει διμερείς συμφωνίες ε, με τις ΕΥΠΑ, οι οποίες δεν είναι και τόσο σωστά κατοχυρωμένες από νομικής πλευράς. Άλλοι δεν έχουν καθόλου τέτοιες συμβάσεις. Ενώ λοιπόν προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε την φόρο διαφυγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνουμε πληροφορίες ε, χωρίς περιορισμού στις ΕΥΠΑ. Έχω ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσβαση σε όλα τα τέτοια δεδομένα που συνδέονται με το ΦΑΤΚΑ την προηγούμενη άνοιξη νομίζω, ακόμα τα περιμένω και θα ήθελα πραγματικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου δώσει αυτά τα έγγραφα και θα ήθελα να καλέσω και αυτή την Επιτροπή και την εισηγήτρια να ε, λάβουν υπόψη αυτό το θέμα. Εάν όχι στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης, τουλάχιστον ξεχωριστά. Very much. Ευχαριστώ κυρία Μέλε. Η κυρία Γκάλς Πέσκ. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια. Συμφωνώ με τα όσα είπε ότι η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή είναι ζήτημα που απαιτεί συντονισμένη δράση. Αυτή τη στιγμή δεν ε, ρυθμίζονται αυτά τα ζητήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να συντονίσουμε τη δράση μα. Κανένα κράτο μέλο μεμονωμένα δεν μπορεί να επιλύσει τα προβλήματα αυτά. Γι' αυτό και η σωστή δημοσιονομική διακυβέρνηση είναι τόσο σημαντική. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την κοινή προσέγγιση. Υπάρχουν, ας πούμε, και αντιστοιχές οδηγίες ε, για τα ε, επιτόκια, για τις πολυεθνικές. Με αυτές τις οδηγίες προσπαθήσαμε να ρυθμίσουμε συγκεκριμένες πτυχές του ζητήματος. Ωστόσο, βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο. Αρκετοί συνάδελφοι είπαν και συμφωνώ ότι ό,τι και αν κάνουμε δεν πρέπει να αυξήσουμε τη γραφειοκρατία. και δεν μπορούμε να δυσκολέψουμε την κατάσταση για όσους συμμορφώνονται με τον νόμο. Επίσης, δεν μπορούμε να περιορίσουμε ε, την, ε, τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Γιατί αυτό θα οδηγήσει σε σημαντικές ε, δυσκολίες. Μπορούμε όμως να βελτιώσουμε τον δημοσιονομικό συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειαζόμαστε βεβαίως τις ε, συναφείς ε, πληροφορίες, ίσως ε, σε έναν ιστότοπο ή μια διαδικτυακή πύλη, όμως αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να γίνεται ταχύτατα. Αλλιώς δεν θα μπορούμε να καταπολεμούμε την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Ένα ενδεχόμενο στοιχείο του νέου πλαισίου θα μπορούσε να είναι η αναθεώρηση των υφιστάμενων μέτρων και της υφιστάμενης νομοθεσίας. Όπως ανέφερε κάποιος συνάδελφος προηγουμένως, και εγώ θα ήθελα να επαναλάβω ότι οι πρακτικές που ακολουθούν όμως υπάρχουν πράγματι διμερείς ε, συμφωνίες για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης, όμως δεν υπάρχει συμφωνία για την διπλή μη φορολόγηση. αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Τώρα, για το σχέδιο δράσης της Επιτροπής, είναι κάτι που έχουμε ήδη θίξει στην Ολομέλεια. Ε, ο μηχανισμός ε, ταχύτατης ανταπόκρισης ε, στην φοροδιαφυγή που αφορά τον ΦΠΑ μέσω αντίστρεφης χρέωσης, αυτός είναι ο μηχανισμός, είναι μια λύση που θα μπορούσαμε να γενικεύσουμε ενδεχομένω. Εγώ θα καταθέσω ορισμένες αντροπολογίες σε αυτό το πνεύμα και θα ήταν πολύ καλό να συνεχίσουμε αυτές τις συζητήσεις με την συγγετρία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μακάρθη. Εντάξει, θα, σύντομα θα είμαι σύντομη γιατί νομίζω ότι και η συγγήτρια ε, μας έδωσε ένα πολύ καλό ε, σχέδιο έκθεσης ε, στο οποίο θα μπορούμε να βασιστούμε για να εργαστούμε. Είναι σημαντικό να μην ξεχάσουμε και το ευρύτερο πλαίσιο. Μόλις τώρα πρόσφατα ετέθη ως προτεραιότητα στη Μόσχα ε, αυτή η ιδέα, πώς δηλαδή θα, θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Παντώντας στις προτάσεις Stretchit, θα πρέπει να είμαστε σαφείς εδώ. Τι προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει ζήτημα δικαιοσύνης. Θα πρέπει δηλαδή να επικεντρωθούμε σε αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές που τείνουν να κάνουν αυτό το forum shopping, να πηγαίνουν δηλαδή όπου τις ε, συμφέρει, χωρίς να τηρούν ε, τις ε, δεσμεύσεις τους. Γι' αυτό και αυτή η ιστορία με τα Starbucks στον Ηνωμένο Βασίλειο, ότι δεν κατέβαλε τους απαραίτητους φόρους στον Ηνωμένο Βασίλειο, οι πολίτες τα μποϊκόταραν τα Starbucks, γιατί είπαν, κοιτά να δεις, εγώ πληρώνω τους φόρους μου, ε, σα πληρώνω για να αγοράσω τον καφέ μου, εσείς γιατί δεν πληρώνετε ε, τους φόρους που σα αναλογούν. Υπάρχει λοιπόν και αυτό το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην ε, φορολογία. Ε, συμφωνώ επίσης με την ιδέα ότι οι μικρές επιχειρήσεις ε, αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα με την εφορία. Αλλά σε ορισμένε περιπτώσει έχω δει αυτή την κατάφορη παραβίαση των ε, κανόνων και βλέπουμε ότι πολλέ φορέ η εφορία κυνηγά του ε, τα μικρά ψάρια ε, με μικρές παραβιάσεις, αλλά δεν έχουν κυνηγήσει ουσιαστικά όσου κατάφορα και κατά συρροή παραβιάζουν τους κανόνες φορολόγησης. Αυτό θα πρέπει να εξετάσουμε επίσης. Είναι το ζήτημα της των χρηματοοικονομικών ε, υπηρεσιών και τον αντίστοιχο κανονισμό. Είδατε προσφάτως ότι η Barclays επιτέλους ε, συμφώνησε καθώς ε, έχει πιαστεί στα πράσα, αν θέλετε, σε περιπτώσεις μεγάλης φοροαποφυγής. Αποφάσισε επιτέλους λοιπόν και συμφώνησε να κλείσει το Tax Efficiency Unit, αυτή τη μονάδα του που ουσιαστικά εργάζεται για να βοηθήσει τους πελάτε να αποφύγουν τη φορολογία. Αυτό κάνουν. Αυτή για μένα είναι η ατζέντα δικαιοσύνης και θα πρέπει λοιπόν να δούμε αν αυτή η βιομηχανία, αυτός ο κλάδος επιχειρήσεων που έχει ε, είχε μεγάλο μερίδιο ευθύνη στην κρίση, έχει αναλάβει το μερίδιο της στην φορολογία. Όλε αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν έχουν ένα τεράστιο αριθμό δικηγόρων και υπαλλήλων με μοναδικό στόχο να βοηθήσουν του πελάτε τους να αποφύγουν ε, την φορολόγηση, να στείλουν τα χρήματά τους σε φοροπαραδείσους για να αποφύγουν τη φορολόγηση. Συμφωνώ με του συναδέλφου με τα όσα είπαν για το ποιε είναι οι ευθύνε μα για τα αναπτυσσόμενε χώρε. αρκετά τέτοια περιστατικά αναφέρθηκαν στον διεθνή τύπο. Ιδίω πριν από δύο εβδομάδε ε, είδαμε ότι από του μεγαλύτερου παραγωγού ζάχαρη, ε, που, ε, στον οποίο νίκη και η εταιρεία Lipton, που είναι και το τσάι που πίνουμε εδώ πέρα, φάνηκε λοιπόν ότι δεν πληρώνει φόρου ε, στην κυβέρνηση τη Ζάμπια. αλλά στέλνει τα χρήματά του σε έναν λογαριασμό στο εξωτερικό και έτσι φόρο αποφεύγει και ταυτόχρονα έχουμε και τη φωτογραφία ενός ε, κοριτσιού που δεν μπορεί να πάει στο σχολείο γιατί δεν ε, υπάρχουν χρήματα να το στείλουν ε, με το λεωφορείο. Ε, υπάρχουν λοιπόν αυτές οι αδικίες και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε γιατί δεν πιάνουμε αυτές τις μεγάλες πολυεθνικές, γιατί δίνεται δυνατότητα σε αυτές τι πολυεθνικές να επιλέγουν ε, χώρες ε, και φορολογικά συστήματα κατά το δοκούν, γιατί καταφέρνουν να μην πληρώνουν τους φόρους που τους αναλογούν, γιατί υπάρχει δυνατότητα να βάλει κάποιο την έδρα τη επιχείρησή του στο Λουξεμβούργο για να πληρώνουν καθόλου φόρους. Επιτέλους λοιπόν αποφάσισαν και συμφώνησαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα ζητήματα ε, οι ηγέτες των χωρών μας ε, στη Μόσχα. Γι' αυτό και εμείς μέσω αυτής της έκθεσης θα πρέπει να τους ε, πιέσουμε γιατί θέλουμε δράσεις και όχι μονολόγια. Και εγώ θα καταθέσω κάποιες τροπολογίες για να σημειωθεί κάποια πρόοδος στην αδικία αυτού του συστήματος ε, που μετακυλεί το βάρος κυρίως ε, στους ε, φορολογουμένους. Ευχαριστώ κυρία Γκουλάχ. Thank you, Pablo. Ευχαριστώ Παύλο. Πολύ σύντομα, γιατί πολλά έχουν υποθεί. Συμφωνώ 100% με το ότι δεν θα πρέπει να βαρύνουμε τις μικρές επιχειρήσεις. Κανένας εδώ στην αίθουσα δεν πιστεύω επίσης ότι δεν έχει εμπειρία με την διαχείριση μιας εταιρείας. Ε, επίσης δεν είναι πρόβλημα με την ε, γραφειοκρατία. Ε, όλες οι εταιρείε, όπως η Google και τα λοιπά, οι οποίες μετακινούνται ας πούμε, δεν έχουν αυτό το πρόβλημα. Ας μην χρησιμοποιούμε αυτές, αυτά τα επιχειρήματα. Ε, βεβαίως δεν πρέπει να βαρύνουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά το πρόβλημα δεν είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη φοροδιαφυγή. Ε, επίσης, στην Ευρωζώνη έχουμε πρόβλημα, αν δεν λαμβάνουμε υπόψη το γεγονός ότι ζητάμε μιλάμε για τα δημόσια χρήματα από τη μία, αλλά από την άλλη δεν κάνουμε τίποτα για τη φορολογία. Θα πρέπει να έχουμε ισορροπημένο λογαριασμό. Αυτό πώς το πετυχαίνεται με τη μείωση των δημοσίων δαπανών ε, και των φόρων. Αυτό είναι παράλογο. Επίσης είναι και θέμα ε, εσωτερικής ενίας αγοράς, όπως είναι και θέμα ισότιμης μεταχείρισης. Και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το επιχείρημα της ε, γραφειοκρατίας, τότε θα έχουμε μια νοοποιημένη αφορολογική βάση. Θα ήταν καλό για τις εταιρείε. Ε, θα ήταν για αυτές, καλό για αυτές που κάνουν ε, α, δουλειές με το εξωτερικό. Συμφωνώ να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα σοβαρά. Εγώ είμαι ισχυρή εισηγήτρια. Συμφωνώ ότι κάνετε καλή δουλειά, κύριε εισηγήτρια. Θέλω να σε ενθαρρύνω να πάτε όμω ακόμα πιο πέρα είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα για να μπορέσουμε να πάρουμε το μέρος μας στους Ευρωπαίους πολίτες. Εάν προχωρήσουμε χωρίς καμία προσπάθεια, κανένα μέτρο για, την, για τα φορολογικά θέματα, σε λίγα χρόνια θα τους χάσουμε τελείως Ευρωπαίους πολίτες από, το, από την πλευρά μας, από το μέρος μας. Ο κ. Στέχο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Συγήτρια, θα μιλήσω φιλανδικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή έχουν τεράστια επίπτωση, χάνονται χρήματα, είναι τεράστια η σημασία για τους πολίτες και για τις οικονομίες των χωρών μας. Και με ανησυχεί πάρα πολύ η στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκαλείται από τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Γι' αυτό λοιπόν χαίρομαι για αυτή την έκθεση ειδικά για όσα λέγονται για τους φορολογικούς παραδείσους. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε αυτά που είπαν πολλοί συνάδελφοι. Ότι βεβαίως πρέπει να αποφύγουμε την γραφειοκρατία. Και βεβαίως η φοροδιαθήκη και η φοροαποφυγή είναι εθνικά θέματα. Δεν μπορούμε εμείς να ρυθμίζουμε υπερβολικά πολύ σε, εθνικό, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί συνήθως οι πιο απλές λύσεις είναι οι καλύτερες. Δεν θέλω να συνδεθεί αυτό το θέμα με το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Δεν νομίζω ότι θα φέρει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Το πιο σημαντικό θέμα στην έκθεσή σας είναι αυτό που λέτε για τους φορολογικούς παραδείσους. Θα πρέπει να συγκρίνουμε τις βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη. Στην ε, Φιλανδία είχαμε σκανδαλώδη παραδείγματα, όπου εταιρείε τα κατάφεραν να αποφύγουν εντελώς τη φορολόγηση. Έγιναν παράσιτα για την κοινωνία αυτές οι εταιρείε. Αντί να είναι πυλώνες κοινωνίας μας. Εν κατακλείδη θα ήθελα να αναπτύξετε περαιτέρω τις ιδέες σας για τους φορολογικούς παραδείσους. Ο κύριος Στρόγιαν, Στρόγιαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας πω μια μικρή ιστορία για το σκάνδαλο του αλογίσιου κρέατος το Μάρτιο στην Ευρώπη. Χαίρομαι που η χώρα μου τη γλίτωσε, γιατί το αλογίσιο κρέας από τη Ρουμανία εστάλει σε άλλες χώρες με νόμιμα έγγραφα, που έλεγαν ξεκάθαρα αλογίσιο κρέας. Κάπου όμως την πορεία, και ενώ ταξίδευε το αλογίσιο κρέας, κάποιος άλλαξε τα στοιχεία, στα έγγραφα και από αλογίσιο κρέας έλεγαν βόλιο κρέας. Αυτό μας το σκάνδαλο έκρυψε μια άλλη ιστορία. Εμένα μου αρέσει να κοιτάω πάντα τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Όταν το κρέας εστάλει από τη Ρουμανία στις διαφορετικές δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, τα έγγραφα ταξίδευσαν προς Ανατολάς. Πρώτα στην Κύπρο και συνεχεία στην Άπο Ανατολή. Όπου εκεί υπήρχε μια άλλη εταιρεία που ήταν μέτοχος μιας ε, κυπριακής εταιρείας και όπου είχε έδρα κάπου στον Ειρηνικό, ούτε και ξέρω εγώ πού. Τι είδους business είναι αυτή. Και για πόσο καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δέχεται τέτοιου τύπου επιχειρήσεις και θα τις θεωρεί νόμιμες. Πίσω από κάθε ε, έγγραφο θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα ελέγχει τα έγγραφα, τις τιμές κτλ. Είναι πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. να κοιτάξει όλους αυτούς τους, να τους ψάξει όλους αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους και να απαιτήσει διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών. Αν αυτή η φορολογική παράδειση δεν δεχτούν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για ανταλλαγή πληροφοριών, για διαφάνεια, θα πρέπει να μπορέσουμε να εμποδίσουμε τέτοιου είδους δραστηριότητες προς αυτούς τους φορολογικούς παραδείσους. Στο παρελθόν ε, πρότεινα ένα πολύ σκληρό μέτρο και δεν συμφωνήθηκε. Καταλαβαίνω γιατί όχι. Γιατί όχι. Θα πρέπει να σταματήσουμε την δραστηριότητα ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που στέλνουν έγγραφα σε τέτοιους φορολογικούς παραδείσους. Εάν αυτοί οι φορολογικοί παράδεισοι δεν συμφωνήσουν να, συνάψουν συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση για διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών. Έχουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη Ρουμανία δισεκατομμυριούχους που δεν πληρώνουν φόρους. Γιατί, Γιατί έχουν τα λεφτά τους σε διάφορες τους παραδείσους, οι οποίοι δεν θέλουν να στείλουν όμως πληροφορίες στις εφορίες της Ρουμανίας για αυτούς τους εκατομμυριούχους ή δισεκατομμυριούχους. Και αυτοί οι δισεκατομμυρίουχοι είναι κάτοικοι για φορολογικούς σκοπούς αυτών των παραδείσων. Δεν θα πρέπει να δεχτούμε αυτές τις συναλλαγές. Έχετε υπόψη σε αυτό το σκάνδαλο του αλογίσιου κρέατος που συνδέεται κιόλα με τέτοιου είδου πρακτικές που χρησιμοποιούν αυτέ οι εταιρείε τέτοιου είδου φορολογικούς παραδείσους Κυκλοφορούν διάφορα έγγραφα, λαθρέα, προς διάφορες κατευθύνσεις και φυσικά δεν πληρώνουν και φόρους αυτές οι εταιρείε. Ευχαριστώ κυρία Στόγιαν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τον λόγο τώρα. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε που μου δίνετε τον λόγο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής σας και τον εισηγητή της εισηγήτρια για το ενδιαφέρον για αυτό το θέμα και το ενδιαφέρον για, όσο, ε, για όλα αυτά τα θέματα που παρακολουθεί. Καλωσορίζουμε το ενδιαφέρον του Ευρωκοινοβουλίου για αυτά τα θέματα. Όπως γνωρίζετε, το ψήφισμα που ενέκρινε το Κοινοβούλιο τον Απρίλιο έχει σημαντική επιρροή σε σχέση με την ε, ε, ενημέρωση που ακολούθησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο και το πρόγραμμα δράσης μας που παρουσιάσαμε το Δεκέμβριο πέρσι. Πολλά θέματα από αυτά που αναφέρονται στο ψήφισμα προσπαθήσαμε να εντάξουμε σε αυτές τις δράσεις. Δύο σημαντικά θέματα είναι εδώ έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το ένα είναι να διασφαλιστούν φορολογικά είσοδα από τα κράτη-μέλη. Από την άλλη πλευρά να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ισοδίκαιο επίπεδο όσον αφορά το σύστημα ίσπραξης εσόδων και την δυνατότητα να συζητηθούν αυτά τα θέματα για να υπάρχει η δικαιοσύνη και αποτελεσματικότητα. Σημαντικό έργο σε αυτό το πλαίσιο. Ως Επιτροπή παρουσιάσαμε το Δεκέμβριο ένα μια δέσμη μέτρων ε, πολύ φιλόδοξη, 34 συνολικά μέτρα, τα οποία όπως ευελπιστούμε θα μπορέσουν να προχωρήσουν τα επόμενα χρόνια έχουν ήδη καθελκιστεί και ξεκινήσει, ιδιαίτερα με συστάσεις που υιοθετήθηκαν ταυτόχρονα όπως και το πρόγραμμα δράσης για την αντιμετώπιση των φοροπαραδείσων και σε σχέση με τις απαιτήσει για τον προγραμματισμό φοροεσόδων πολλές ιδέες από αυτές που εκφράστηκαν σήμερα σε αυτή τη συζήτηση και θα ε, καλωσορίζαμε την υποστήριξη από το Ευρωκοινοβούλιο των δικών μας αυτών πρωτοβουλειών. Με τη δική σας υποστήριξη θα είμαστε σε πολύ ενδυναμωμένη θέση ώστε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να αναλάβουν κοινή δράση επ' αυτών των θεμάτων. Ευχαριστώ Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τέλος θα δώσουμε τον λόγο στην εισηγήτρια και πάλι. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ. Τις παρατηρήσεις ε, κλείδι θα τις κάνω στα σλοβενικά στη μητρική μου γλώσσα και θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και αυτή τη γλώσσα. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να ξεκινήσω λέγοντας ότι ευχαριστώ σου συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση και ευχαριστώ για τις προτάσεις σας. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι βέβαια καινούριο. Συζητήσαμε και συζητούσαμε αυτό το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο για αρκετό χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα σε αυτήν την Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η κύρια ιδέα σε σχέση με αυτή την έκθεση και ξέρετε πόσο ποιοι περιορισμοί είναι δεδομένοι για τη σύνταξη τέτοιων εκθέσεων, είναι μια έκθεση που θα ενδυναμωθεί και θα βελτιωθεί πρέπει να πω και θα τροποποιηθεί και θα προσαρμοστεί ανάλογα με τις τροπολογίες που ε, καταθέτουν τα μέλη εσείς και προσβλέπω λοιπόν σε αυτές τις τροπολογίες ώστε να τις εξετάσω και να δω τι μπορούμε να κάνουμε. Από κοινού πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να είμαστε σε θέση να καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα είναι υπερήφανο το Ευρωκοινοβούλιο να παρουσιάσει στους ε, ηγέτες των κρατών μελών ε, που συζητούν και ασχολούνται με αυτά τα θέματα και τους απασχολούν στην λέσχη των 20 για παράδειγμα G20 όπου Κάποιες υποσχέσεις ε, δίνονται που στη συνέχεια όμως ε, δεν μεταφράζονται σε συγκεκριμένες χειροπιαστές δράσεις. Ελπίζω ότι η έκθεση θα έχει επιπτώσεις λοιπόν στα όσα τεκταίνονται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όσον αφορά την, ε, τα θέματα αυτά, η Επιτροπή Ανάπτυξης προετοιμάζει ένα συγκεκριμένο έγγραφο και συμφωνήσαμε να κατανείμουμε, να επιμερίσουμε το έργο μεταξύ μας. Είμαι, έχω την βεβαιότητα ότι θα κάνει εξαιρετική δουλειά η Επιτροπή η Επιτροπή Απασχόλησης. Σε σχέση με τα όσα προανέφερα, αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Ήθελα να δείξω ποια είναι τα κονδύλια τα οποία στο τέλος τέλος χάνονται και η απώλειά τους λόγω φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής καταλήγει σε αυτή την κατάσταση. Είναι μια κατεκτήμηση λοιπόν παρουσίαση της κατάστασης και αφορά τα αριθμητικά μεγέθη που ε, δόθηκαν. Ορισμοί. Τώρα για τους ορισμούς ε, είναι πραγματικά ε, επώδυνο το θέμα. Θα ήθελα να μπορούσαμε να καθορίσουμε στο τέλος το πρόβλημα των φοροπαραδείσων με ένα πιο συντονισμένο τρόπο δεν καταφέραμε να το κάνουμε αυτό μέχρι σήμερα. Αν τα καταφέρουμε όμως, αν μπορέσουμε να είμαστε επιτυχείς και καταλήξουμε σε έναν αποτελεσματικό ορισμό σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή στην Ευρωβουλή μας θα το δεχθώ με μεγάλη ικανοποίηση. Σε όλες τις συζητήσεις και διαβουλεύσεις που είχα μου είπαν οι εμπλεκόμενοι μη δώσετε συνέχεια σε αυτό είναι υπερβολικά δυσχερές το εγχείρημα όμως παρόλα αυτά αποφάσισα να δώσω συνέχεια και να προχωρήσω το αποτέλεσμα της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Όλα αυτά τα θέματα πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, ώστε να κερδίσουμε στο τέλος ως αποτέλεσμα την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών μας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και από πλευρά των επιχειρήσεων να υπάρχει ένα αποτελεσματικό ισοδίκαιο δίκαιο σύστημα και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε αυτή την έκθεση με τις τροπολογίες σας και προτάσεις σας. Ελπίζω ότι θα μπορέσει να γίνει πιο αποτελεσματική και συγκεκριμένη η έκθεση έχω κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις από πλευράς μου που συμπεριέλαβα στις διατυπώσεις μου, αλλά έχω τη βεβαιότητα ότι θα υπάρξει επαρκής χρόνος να βελτιωθεί περαιτέρω η έκθεση. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και ευελπιστώ ότι θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία. Πρόεδρος, υπενθυμίζω ότι 26 Φεβρουαρίου είναι ε, η ημερομηνία κατά την οποία η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Στις 20 Μαρτίου θα εξετάσουμε και η ψήφιση θα γίνει στις 24 Απριλίου και στο τέλο η θα περάσουμε στην Ολομέλεια ώστε στην περίοδο συνόδου του Μαΐου να διεκπαιρεωθεί το θέμα. Περνάμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, το θέμα 15. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης ε, όσον αφορά την, ε, τα προβλήματα συνταγματικής φύσης σε μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συγγήτρια είναι η κυρία Σιλβί Γκουλάρ. Έχετε τον λόγο κυρία Γκουλάρ. Ευχαριστώ είναι ένα αρχαιολογική ανασκαφή σχεδόν αυτό που σας προτείνω να κάνουμε σήμερα, γιατί η ιδέα αυτή της έκθεσης είχε ξεκινήσει πριν από ένα χρόνο περίπου, ίσω και παραπάνω, σε μια χρονική στιγμή που ακόμα δεν υπήρχε αυτό το εγχείρημα του κυρίου Βαν Ρόμποϊ, δεν υπήρχε η έκθεση Βαν Τάισεν κτλ. κτλ. Έχουμε λοιπόν ένα κείμενο που έχει μείνει στο σιρτάρι, αν θέλετε, και Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι καλό η Επιτροπή μας ε, να εκφέρει γνώμη. Είναι σημαντικό το ζήτημα, αφορά την Επιτροπή μας, γιατί προφανώς ό,τι αφορά τη διαφοροποίηση των διαφόρων επιπέδων ε, και σε ό,τι αφορά και τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την Ευρωζώνη είναι εξαιρετικά σημαντικό. Προσπάθησα λοιπόν ε, να ε, αντιμετωπίσω αυτό το θέμα ως εξής. Ε, να υπερασπιστώ τις αρμοδιότητες ε, της εικόν σε ό,τι αφορά τις δικές μας ενέργειες και να μην βεβαίως υπησέλθω στις αρμοδιότητες της ΑΦΚΟ και είναι ένα εξαιρετικά σύντομο κείμενο. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι αντί να μπούμε μέσα σε ένα κύκλο αντιθέσεων και διαφορών, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει μια τέτοια, ε, ε ένας διαχωρισμός, ένας διχασμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, ούτως ώστε τα, οι χώρες της Ευρωζώνης και όλες οι χώρες που θα προσχωρήσουν σε αυτή, χώρες δηλαδή που έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη. Θα πρέπει λοιπόν όλε αυτές τις χώρες να ε, συνεργαστούν και να συντονιστούν όσο το δυνατόν καλύτερα, ξεκινώντα και από αυτή την ε, λογοδοσία που απαιτείται, ε, παρά τι δυσκολίε της κρίσης και χωρίς να υπάρχει αυτό ο διαχωρισμό. Βεβαίω λοιπόν... Αναφέρθηκε ότι υπήρξε μια δημοσιονομική εξυγίανση και αυτό είναι ικανοποιητικό. Υπήρξε μηχανισμός αλληλεγγύης που δεν υπήρχε προηγουμένως. Ε, αναφερθήκαμε στην ύπαρξη της Τρόικας που πάει σε ορισμένες χώρες χωρίς να αναφερθούμε στον τρόπο ε, εργασίας της. Μετά για τις πρόνοιες που υπάρχουν και τι διατάξεις που υπάρχουν για να διασφαλίζεται ότι αυτέ οι χώρες ε, τηρούν τι δεσμεύσει του και ούτω καθεξής. Ε, αυτά εν ολίγης, ε, είμαι ανοιχτή σε προτάσει. Και βεβαίως πρέπει βασικό μας μέλημα να είναι ένα πολύ συγκεκριμένο μήνυμα προς την Επιτροπή ΑΦΚΟ ότι αρκετά πράγματα έχουν γίνει και στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων κάτι το οποίο αιτιολογεί μια τέτοια εξέταση χωρίς να υπάρχει ούτε διαχωρισμός ούτε διχόνοια, χωρίς όμως να ελαχιστοποιούμε και να ε, παραβλέπουμε και το πιο ουσιαστικό βήμα των κρατών μελών τα τελευταία χρόνια, που ήταν δηλαδή η απόφασή να συμμετάσχουν ή όχι στην Ευρωζώνη. Και μέσα στα και στα επόμενα σημεία αναφέρω και του, τον, την ευθύνη μας απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες και μετά μιλάω για την Ένωση και όχι μόνο για έναν αριθμό κρατών μελών και η ίδια ε, η συνθήκη αναφέρει ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι προσωρινά γιατί όλοι θα προσχωρήσουν κάποια στιγμή στην Νομισματική Ένωση. Επομένως, θα πρέπει ακόμα παραπάνω να εξετάσουμε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Γκουλάχ, ο κύριος Ρωσές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Σιλβή καλά λέει ότι πρόκειται για αρχαιολογική ανασκαφή, γιατί εμένα μου είχε ξεφύγει αυτή η ε, έκθεση και πράγματι πρέπει να τρέξουμε στο μακρινό παρελθόν για να βρούμε τις απαρχές της έκθεσης. Ε, εγώ με σκιώδης συζητής, δεν είναι πρώτη φορά. Ήθελα μόνο να πω ότι επί της προσέγγισης συμφωνούμε. Ε, μια μικρή παρατήρηση για το σημείο 5, γιατί στο γαλλικό ε, μιλάμε για ε, λεπτομερές σχέδιο και όχι blueprint που είναι ο αρχικός αγγλικός ε, όρος. Πολλές φορές αφορά χρηματοοικονομικά ζητήματα το blueprint. Αναφερόμαστε λοιπόν στις προσπάθειες της Επιτροπής, που όμως δεν έχει όμως αποτελέσει ακόμα ε, αντικείμενο διεξοδικής συζήτησης. Αυτή είναι η μόνη μικρή παρατήρηση που έχω να κάνω. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε με τα όσα μόλις είπες. Γιατί το ευρώ αυτή τη στιγμή θα είναι ε, το ε, νόμισμα ολόκληρης Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, επομένως θα πρέπει να έχουμε και συμπεράσματα από θεσμικής πλευράς και να μην διατηρήσουμε αυτή την αρχή που υπάρχει σήμερα ότι όλοι ασχολούνται με το ευρώ επειδή το ευρώ έχει ως σκοπό να γίνει το νόμισμα όλων. Και αν αυτό δεν ισχύει, τότε θα πρέπει να υπάρχουν και οι απαραίτητες θεσμικές ε, ε, επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκρόσες. Για τους σοσιαλιστές, να δώσω το λόγο στον κύριο Κούρτας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της, για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης και να αναφέρω ότι αρκετές ε, μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να πραγματοποιηθούν για την πιο εύρυθμη λειτουργία της ε, Νομισματικής Ένωσης και για την ενίσχυση ε, του δημοκρατικού ελέγχου. Συμφωνώ με την πρόταση σε ό,τι αφορά με την Τρόικα και τους ιδίους πόρους και για τους ιδίους πόρους επίσης και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η ε, ε, ανάγκη δημιουργίας ε, ευρωπαϊκού θησαυροφυλακίου, αν θέλετε, Υπουργείου Οικονομικών. Και ο δικός μας ρόλος βεβαίως ως Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο είναι εξαιρετικά σημαντικός εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το Κοινοβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι το ε, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πολύ σωστά εκπροσωπεί και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ΟΝΕ. Όπως ξέρετε, δύο συνάδελφοι στην Επιτροπή ε, Συνταγματικών Υποθέσεων ε, ανέφεραν ότι η εγκυρότητα του Six ποτέ δεν αμφισβητήθηκε, παρότι έχει ψηφιστεί και από τα μέλη της Ευρυζώνης και από τα κράτη-μέλη που δεν είναι μέλη της Ευρωζώνης. Αυτή η συζήτηση μεταξύ ε, μελών της Ευρωζώνης και μελών που δεν είναι στην Ευρωζώνη μπορεί να ανοίξει το κουτί της Πανδώρας ε, και να έχει επικίνδυνες για ζητήματα σταγματικής φύσης σύμφωνα με ορισμένα άρθρα του, της συνθήκης του 10 και του 14 η Ευρωπαϊκή Ένωση εκπροσωπεί όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και έτσι λοιπόν εμείς θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτά τα στοιχεία και όχι να τα αποδυναμώσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Από τους πράσινους. Ευχαριστώ. Σάικο. Ευχαριστώ Σιλβία για την καλή έκθεση. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη από τον Ζαν Πολ Γκοζές που ζήτησε να δώσει τη γνώμη του για αυτό το θέμα, ενώ κανονικά έπρεπε να βρίσκεται σε μια άλλη ψηφοφορία, σε μια άλλη επιτροπή. Ευχαριστώ για τη βάση αυτής της έκθεσης. Σε μεγάλο βαθμό συμμερίζομαι αυτή τη βάση. Το μόνο που θέλουν να πούν οι πράσινοι είναι ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε την έκθεση σε κάποια επιμέρους σημεία, όπως είπατε και εσείς, έχετε περιορισμό λέξεων και χώρου. Εντάξει, θα το λάβουμε υπόψη μας. Θα πρέπει παρόλα αυτά να ενισχύσουμε κάποια σημεία. Κάτι που πρέπει να πούμε είναι ότι τελικά ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ε, πρέπει να λειτουργήσει με την κοινωτική μέθοδο για την Τραπεζική ε, Ένωση. Ε, το ενιαίο σχήμα εγγύηση των καταθέσεων και ο ενιαίος μηχανισμός ε, εποπτείας θα πρέπει να είναι βασικοί πυλώνες. Για τις διμερείς συμφωνίες που αναφέρονται και θα συζητηθούν ε, στο Συμβούλιο ξανά του Ιουνίου, από πλευράς Κοινοβουλίου θέλουμε να πούμε ότι αυτές οι διμερείς ε, συμφωνίες θα πρέπει να την χάνουν δημοκρατικής λογοδοσίας και απολογισμού και επιπλέον αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να τις ημερίζονται και οι διάφοροι φορείς σε εθνικό επίπεδο και αν τις εγκολπώνονται. Ε, το άρθρο που μιλάει για τους ίδιους πόρους, τέλος πάντων. Θέλω να σας πω ότι στην τελική βα... ε, οι πόροι είναι η βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσουμε και τα σύμμετρα σοκ. Αυτά είναι κάποια από τα σημεία που θέλουμε να προσθεθούν στην έκθεσή σας, Σιλβή. αλλά σε ευχαριστώ ακόμα μια φορά ξανά και ξέρω ότι ο Ζων Πολ ε, θέλει με μεγάλη ανυπομονησία να συνεργαστεί μαζί σας. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα από την ε, ECR, ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τρία σχόλια θέλω να κάνω. Στην παράγραφο 2 του σχεδίου γνωμοδότησης, η κυρία Γκουλάρ λέει ότι το six-pack αφορά μόνο τα μέλη της Ευρωζώνης. Δεν ισχύει νομίζω αυτό. Το six-pack αφορά και τα 27 κράτη-μέλη. Παρότι κάποιοι κανόνες σε ό,τι αφορά τις ε, οικονομικές κυρώσεις αφορούν ειδικά τα μέλη της Ευρωζώνης. Επομένως, θα ήθελα να, γίνει, να δοθεί κάποια διευκρίνηση εδώ, αν μπορεί η κυρία Γκουλάχ. Το 2 αφορά αποκλειστικά τα μέλη της Ευρωζώνης. Θέλω να υπενθυμίσω στην Επιτροπή σας ότι η πολιτική ομάδα της κυρίας Γκουλάρ ε, μπλοκάρει την υιοθέτηση αυτού του πακέτου που το χρειαζόμαστε τα μάλα. Επίσης, στην παράγραφο 5 του σχεδίου γνωμοδότησή της, η κυρία Γκουλάρ ζητά να υπάρξουν νέες νομοθετικές προτάσεις. Θέλει να εφαρμόσει το blueprint της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παράγραφο 7 λέει ότι η Ευρωζώνη χρειάζεται ξεχωριστό προπολογισμό. Είπα ξανά ότι η Ευρωζώνη δεν θα πρέπει να γίνει μια οικονομία μεταφοράς. Θα πρέπει να βασίζεται σε βάση καθαρούς κανόνες, δημοσιονομική πειθαρχία και κυρώσεις για αυτούς που παροβιάζουν τους κανόνες αυτούς. Αυτό είναι το πνεύμα του Μάστριχτ και θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπάθουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Στην παράγραφο 8 η κυρία Γκουλάρ επίσης ζητάει την εισαγωγή ενός κοινοβουλίου της Ευρωζώνης. Ακόμα ένα ε, κοινοβούλιο δηλαδή. Θέλει μια, ένα υποσώμα ε, του κοινοβουλίου που θα απαρτίζεται από τα μέλη της Ευρωζώνης ή από μέλη που δεν ανήκουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη, που θα ενταχθούν στο μέλλον. Εμείς τι είμαστε τότε. Ε, θα έχετε την ίδια προσέγγιση, κυρία Συγγήτρια, και για το Σέγγεν. Θα δημιουργήσετε ένα κοινοβούλιο για το Σέγγεν και για κάθε ε, τομέα ενισχυμένη συνεργασία θέλετε ειδικό κοινοβούλιο. Δηλαδή, όπω παραδείγματο χάρη ένα κοινοβούλιο πούμε, για το φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών. Καταλαβαίνω γιατί τα προτείνετε αυτά που προτείνετε. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε τελικά. Ότι θέλετε ένα κοινοβούλιο χωρίς μέλη από το Ηνωμένο Βασίλειο. Παρότι εγώ εκπροσωπώ το Βέλγιο, έτσι δεν είμαι από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν θέλω τέτοιου τύπου ιδέες. Και θα πρέπει ακριβώς για το καλό των πολιτών, τους οποίους επικαλείστε τόσο συχνά, να αποφύγετε αυτά, τα, αυτόν τον κατακαιρματισμό της κοινοβουλευτικής εποπτείας. Λοιπόν, η Γκουε δεν θέλει νομίζω το λόγο γιατί δεν έχει κανένα μέλο εδώ. Ο κύριο Τρεμόζα ζητάει το λόγο. Θα το δώσω. Ένα λεπτό. Σε ένα λεπτό να πω ότι σε σχέση με την χρηστή ε, διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση με χαρά διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα στο περιοδικό Economist το άρθρο ε, Charlemagne όπου αναφέρθηκε και το σχετικό για το Ευρωκοινοβούλιο που είναι ένα κοινοβούλιο που υπάρχει εκπροσώπηση χωρίς όμως φορολογικά δικαιώματα επιβολής φόρων. Και αυτό είναι το θέμα που έχει τη μεγαλύτερη σπουδαιότητα. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το εγχείρημα πρέπει να αντιληφθούμε ότι θα υπάρχει ε, πρόβλημα. Θα πρέπει να αποφασίσουμε να περάσουμε στο επόμενο βήμα, στην επόμενη κλίμακα, δηλαδή οι φορολογικές αρμοδιότητες. Δεν θα είναι δική μας η απόφαση, θα ληφθεί από τους Ευρωπαίους πολίτες ε, που ε, στις επόμενες εκλογές θα πρέπει να τοποθετηθούν. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το θέμα και θα δούμε πόσο σπουδαίο, πόσο σημαντικό είναι. Κάνοντας λόγο επίσης από την άλλη πλευρά για την ενδυνάμωση της ε, σταθερότητας, της αποτελεσματικότητας και της δημοκρατικής λογοδοσίας, θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη ότι θα πρέπει να γίνει λόγος εξίσου ότι υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι αρκετά αποτελεσματικά στις επιδόσεις τους ε, εφόλων αυτών. Και τώρα σε σχέση με την αρχή ε, δεν θα υπάρχει φορολόγηση χωρίς εκπροσώπηση ή αντίστροφα δεν θα υπάρχει εκπροσώπηση χωρίς φορολόγηση, πρέπει να ζητηθεί να υπάρξει φεντεραλισμό ε, φορολογικός ε, σε σχέση με τις μεγάλες ε, χώρες της Ευρώπης, όπως π.χ. και στην Ισπανία Ολοκληρώνοντας αυτή την ιδέα ως προοπτική, αν εξετάσουμε την εξέλιξη της ευρωπαϊκής οικονομίας τα τελευταία πέντε χρόνια με αυτή την τεράστια οικονομική κρίση, οι καλύτερες τις επιδόσεις τους χώρες, τα καλύτερα κράτη τις επιδόσεις τους, επειδή μπόρεσαν να βρουν άμεσα λύσεις, είναι οι μικρές χώρες της ε, Σκανδιναβίας, της Βόρειας Ευρώπης και η Γερμανία ως εξαίρεση λειτουργεί ως σκανδιναβική χώρα σε αυτό το πλαίσιο, διότι είναι μια αυθεντική ομοσπονδιακή χώρα στη δομή της. Υπάρχουν 17 κρατήδια που έχουν εξουσίες πλήρους φορολόγησης από πλευρά τους και έχουν και εξουσιοδότηση να προβαίνουν στη ρύθμιση των θεμάτων υποδομών, για παράδειγμα σιδηροδρόμων, αερολιμένων κτλ. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι η επιδόσεις, η αποτελεσματικότητα συνδέεται και με τις διαστάσεις και η καλύτερη ευρωπαϊκή απάντηση δόθηκε από τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, τις σκανδιναβικές χώρες. Γιατί υπάρχουν προβλήματα στην Ιταλία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, ίσως και στη Γαλλία ακόμα και στο Βέλιο δηλαδή ε, στις νοτιότερες χώρες της Ευρώπης. Επειδή υπάρχει μόνο μία κεντροποιημένη κρατική δομή ως ε, μία υπηρεσία και ε, σε αυτήν εντάσσονται όλες οι άλλες εξουσίες, υποδομές κτλ. Όταν κάνουμε λόγο λοιπόν για την διακυβέρνηση επαυτών στην Ευρώπη, ζητούμε να υπάρχει αποτελεσματικότητα, δημοκρατική λογοδοσία, ενδυνάμωση της σταθερότητας. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να κάνουν τα του οίκου της, να κάνουν σωστά τη δουλειά του. Δεν γίνεται να συζητούμε ε, για τους ιδίους πόρους στο ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς να λάβουμε καθόλου υπόψη αυτά τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν από πλευρά κρατών μελών. Ευχαριστώ, Πρόεδρο, σας ευχαριστώ αγαπητέ Ραμόν, όχι μόνο χρειαζόμαστε αποτελεσματικά πολιτικά συστήματα. Χρειαζόμαστε και καλές ε, χρηστές κυβερνήσεις για την χρηστή διακυβέρνηση. Γκουλάρ παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ Παύλο, σας ευχαριστώ όλους. Με μεγάλη χαρά άκουσα ότι ο Ζωάν Πολ και άλλοι μπορούν να με βοηθήσουν. Όλοι και αυτοί που πήραν τον λόγο και όσοι είναι απόντες. Επίσης, μπορούμε να επιμηκύνουμε το, το κείμενο. Κανένα πρόβλημα αλλά υπάρχει όμως ε, όριο λέξεων αυστηρό. Ε, να πω στον συνάδελφο εδώ στα δεξιά μου. Λαμβάνω υπόψη αυτό που λέτε για, για τα, τις χώρες μέλη του ευρώ. Και συμφωνώ με αυτό που είπε ο κ. Κούτας, ότι δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα άλλο κοινοβούλιο. Αντίθετα, Θέλουμε μεγαλύτερη ευελιξία στο εσωτερικό του υπάρχοντος κοινοβουλίου, ούτω ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε αποφάσεις με σχηματισμούς που δεν θα αποκλείουν κανένα, που θα επιτρέπουν σε όλους τους συναδέλφους, αν δεν ανήκουν, να είναι παρατηρητές και αν ξαφνικά μια χώρα αλλάξει καθεστώς και πάει από το ένα στρατόπεδο στο άλλο, μπορεί να αλλάξουμε κι εμείς σχηματισμό αν εμεί ω Κοινοβούλιο δεν λάβουμε υπόψη μα το αίτημα που υπάρχει από τους ευρωπαϊκούς πληθυσμού να κάνουμε τα πράγματα με απλό τρόπο, δηλαδή το να συμμετέχουν σε μια απόφαση αυτοί που αποφάσισαν κυριαρχικά να συμμετάσχουν σε ένα project ας πούμε και να μην τιμωρήσουμε τους άλλου που αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν. Όλα αυτά καλά να είναι να τα κάνουμε στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Αν το Κοινοβούλιο δεν συνειδητοποιήσει ότι θα πρέπει και αυτό να επιδείξει ευελιξία, ε, ο κίνδυνο ποιο είναι. Να δημιουργήσουμε δομέ οι οποίε εκφεύγουν του κοινοτικού ελέγχου. Αυτό ε, έγινε ε, με την δημοσιονομική συνθήκη, με το ESM κτλ. Έχουμε πολλαπλασιασμό των δομών που εκφεύγουν αυτού του ελέγχου. Και αν είναι εκτό, ε, τα πράγματα είναι ακόμα πιο σοβαρά. Γιατί εδώ τουλάχιστον έχουμε την δυνατότητα να δώσουμε, να προσφύγουμε και να βρούμε λύσεις προσωρινού χαρακτήρα, να λειτουργήσουμε με ευελιξία κτλ. Επίσης, είμαι ανοιχτή σε κάθε πρόταση αλλαγής που θα μας επιτρέπει να λάβουμε υπόψη όχι αυτό που ήταν μέχρι στιγμής η ορθοδοξία του Κοινοβουλίου και των συνθήκων, αλλά να απαντήσουμε στις θεμητές προσδοκίες των πληθυσμών μας και που αν τις αγνοήσουμε θα λυθούν υπόψη από τα κράτη-μέλη μέσα σε ένα πνεύμα διακυβερνητικό και από αυτό δεν έχουμε να κερδίσουμε σε καμία περίπτωση. Ευχαριστώ Σιλβί. Τελειώνουμε εδώ τη συζήτηση και σας υπενθυμίσω ότι στις 19 Φεβρουαρίου θα συζητήσουμε την έκθεση. Η προθεσμία για τις τροπολογίε είναι 25 Φεβρουαρίου. Ε, θα εξετάσουμε τις απολογίες στην Επιτροπή στις 11 Μαρτίου και η ψηφοφορία στην Επιτροπή ΕΚΟΝ θα λάβει χώρα στις 21 Μαρτίου, στην καθήλυνα αρμόδια Επιτροπή ΑΦΚΟ στις 23 ε, Μαρτίου και δεν ξέρουμε ακόμα πότε θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. 16. Τα διάφορα. Δεν έχουμε τίποτα. Στο 17 ε, είναι η επόμενη συνεδρίαση που θα γίνει την επόμενη Δευτέρα 25 από τις 3 έως τις 6.30 το απόγευμα και την Τρίτη την επόμενη μέρα από τις 9 μέχρι τις 12.30. Σας ευχαριστώ όλους. Υπότιτλοι